Dear uh, good morning. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρωινή συνεδρίαση. Μετά από την ε, φορτωμένη μέρα χθες ε, που συναντηθήκαμε με υπουργούς ε, από την Κροατική Προεδρία και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κυρία Βεστάρ και μετά από μια πολύ φορτωμένη μερίσια διάταξη φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Ε, για μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε για δεύτερη φορά στην Επιτροπή μας, μετά την ακρόασή της, την Επίτροπο Ενέργειας, κυρία Κάντρι Σίμψον. Και όπως γνωρίζετε στις 10.30 θα ακολουθήσει ακρόαση σχετικά με το ορίζον Ευρώπη και την ερευνητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα όμως θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Σίμψον, η οποία δέχτηκε την πρόσκληση να έρθει στην Επιτροπή μας, ε, προς μεγάλη μας χαρά. Θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο. στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας που έχουμε συζητήσει ήδη αρκετά θα εξετάσουμε θέματα ενεργειακής πολιτικής που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Θέματα ενέργειας και όχι μόνο. Φυσικά, τον Ιανουάριο παρουσιάστηκε και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που είναι πολύ σημαντικό θέμα για εμάς, όπως είδατε κιόλας από αυτές τις μέρες. Και επίσης προτάσεις για κλιματική ουδετερότητα, πρόταση αύξησης 50% των στόχων μας μέχρι το 2030, ε, ανακαινήσεις, ε, αναθεωρήσεις του κανονισμού για την ενέργεια και για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θα γίνει σήμερα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σίμψον για 10 λεπτά και στη συνέχεια όπως ε, κάνουμε συνήθως θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος ε, ερωτήσεων από τους συντονιστές. Ε, μέχρι τρία λεπτά ο καθένας σας έχει χρόνο Απίτα η κυρία Σίμψον θα απαντήσει. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο γύρος ερωτήσεων, όπου όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν ερωτήσει. Θα σα παρακαλέσω να δείξετε ότι θέλετε να λάβετε το λόγο τον νωρίτερο. Και στη συνέχεια φυσικά η κυρία Σίμψον θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Και θα κάνει τα καταληκτικά της σχόλια. Περνώ ευθύ αμέσω στην κυρία Πίτροπο. Γνωρίζω πως όλοι περιμένατε να την ακούσετε. Έχετε λοιπόν το λόγο κυρία Σίμψον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας για να σας παρουσιάσω τις ε, κύριες κατευθύνσεις της ε, Πράσινη Συμφωνία από οπτική γωνία τη ενεργειακή πολιτική. Η πρόεδρο Φοντερ Λάιεν είπε ευθύ αμέσω ότι η Πράσινη Συμφωνία θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της νέας επιτροπής και θα πρέπει να αλλάξει δραστικά ο τρόπος ε, λειτουργίας και σκέψης μας, να γίνει μια θεμελιώδης ε, μετάβαση προς ε, μια οικονομία ουδέτερη ως προς τον άνθρακα που συνεπάγεται μείωση των εκπομπών. Οι εκπομπές του ενεργειακού τομέα αποτελούν το 75% των συνολικών εκπομπών αερίου των θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν μια συντονισμένη κοινή προσπάθεια για να αλλάξει αυτό, το οποίο είναι προϋπόθεση ε, για την αποδέσμευση από άνθρακα και των υπόλοιπων τομέων. Το ψήφισμα για την Πράσινη Συμφωνία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα δείγμα της δέσμευσης που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τηρήσει την Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ε, προκλήσεις που έχουμε ενωπιών μας. Έχει στόχο να αποδεσμεύσει την ανάπτυξη από, τους, ε, από τις πρώτες ύλες. Έχει στόχο να εξυγχρονίσει και να μειώσει τον περιβαλλοντικό ε, αντίκτυπο της ενέργειας στην οικονομία μας. Η αλλαγή αυτή σημαίνει πως ορισμένοι τομείς ε, θα έχουν μεγαλύτερες προκλήσεις από άλλους. Αυτό το αναγνωρίζουμε και προσπαθούμε να είμαστε προορατικοί έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση για όλες τις ε, γεωγραφικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει το, ε, τον μηχανισμό δίκαιης προσαρμογής και ένα συνοδευτικό επενδυτικό σχέδιο. Στην ε, Ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας συζητήσατε και εσείς το θέμα, ε, αλλά θα ήθελα και εγώ να σας ε, παρουσιάσω ορισμένε πτυχές του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, οι οποίες μου είναι πολύ σημαντικές. Καταρχάς, είναι ένα ε, ταμείο που θα έχει στόχο να αντιμετωπίσει ε, το δύσκολο έργο της μετάβασης ε, προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Θα συνοδεύεται από διάφορες πρωτοβουλίες και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες χρειάζονται επενδύσεις, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να καταρτιστεί ξανά και χρειάζονται πλατφόρμες μετάβασης. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων. Τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν και αυτά με τα δικά τους εθνικά σχέδια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτάσεις που ε, παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Green Deal και της νέας ενεργειακής πολιτικής. Πρώτον, ε, η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ζωτική σημασία για τη μετάβαση προ καθαρή ενέργεια. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε να, φροντι... να υλοποιηθεί. Έπειτα θα συνοδεύσουμε ε, τη... τα σχέδια των κρατών μελών με συγκεκριμένε κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα επίπεδα πολιτικής. Και για ε, την αρχή το προφανές είναι να δώσουμε έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Αυτό φυσικά από μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζεται να πυροδοτήσουμε ένα κύμα ανακαινήσεων γενικότερο έτσι ώστε να γίνει σε μεγάλη κλίμακα. Χρειάζεται συντονισμένη δράση βέβαια ε, και σε τοπικό επίπεδο από τους πολίτες, από τους υπεύθυνους πολιτικής και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πρωτοβουλία για τις ανακαινήσεις θα συμπεριλάβει και την ε, κοινωνική στέγαση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, και το θέμα των, της ευτόχειας. Θα ασχοληθούμε επίσης και με τα σχολεία, διότι τα τελευταία νούμερα που έχουμε μας δείχνουν ότι το 50% των ε, κτηρίων και των σχολείων δεν έχουν τη δυνατότητα θέρμανσης. Έπειτα, η ενεργειακή αποδοτικότητα των ηλεκτρικών οικιακών ε, συσκευών είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα υπάρξει ένα ε, αντίστοιχο πρόγραμμα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συσκευών και να χρησιμοποιήσουμε την κυκλική οικονομία. Επίσης, ε, η ψήξη και θέρμανση μέσω του ηλεκτρισμού ε, και η χρήση του ηλεκτρισμού στις μεταφορές σκοπεύουμε να γίνει πιο αποδοτική χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος είναι να, μειωθεί, να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος οικονομικά και αυτό θα γίνει μόνο με τη δημιουργία ευφυών συστημάτων που θα χρησιμοποιούν μεν ε, την ηλεκτρική ενέργεια αλλά ε, θα στηρίζονται εν μέρη και ε, στο φυσικό αέριο το 31% της ηλεκτρικής ενέργειας ε, που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχει πολύ χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Το φυσικό αέριο επίσης αποτελεί το 1 τέταρτο της ε, συνολικής ποσότητας ενέργειας στην Ευρώπη και αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ποσοστό. Βέβαια, η μετάβαση προς το φυσικό αέριο θα εξαρτηθεί από τις πρωτοβουλίες του κάθε κράτους μέλους και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες για καθαρό φυσικό αέριο. Και στην αυτοκινητοβιομηχανία το φυσικό αέριο θα διδερματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάζονται οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής αγοράς της Ένωσης, ιδιαίτερα στην ε, περίπτωση ανάπτυξης ε, μεγάλων δικτύων ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας. Ο στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και καθαρή ενέργεια είναι ένα βασικό στόχο τη επιτροπή. και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τις ενεργειακές υποδομές. Θα παρουσιαστεί ε, αντίστοιχη πρόταση μέχρι το τέλος του 2020, όπου θα τονίζεται η χρήση της ε, πρωτοπόρου και καινοτόμου τεχνολογίας όπως ε, τα δίκτυα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, ε, χρήσης ε, υδρογόνου κτλ. Η πολιτική υποδομών χρειάζεται να είναι προστατευμένη από μελλοντικέ προκλήσεις και να φροντίσουμε έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Θα στηρίξουμε λοιπόν διάφορα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας σε υπεράκτιες ε, πλατφόρμες με τη χρήση αιωλικής ενέργειας και άλλα συνοδευτικά μέτρα όπως διαχείριση χώρου, βιομηχανική πολιτική κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς ε, σήμερα και πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την ήδη ισχυρή θέση. Η έρευνα και η καινοτομία τώρα είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία του εγχειρήματο και χρειάζεται να φροντίσουμε έτσι ώστε το κόστος ε, να μειωθεί να, να υπάρχουν λύσεις προσιτές στην αγορά και να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες καλές οικονομικές προοπτικές για την καθαρή ενέργεια. Αξιότιμα μέλη. Για να γίνει πραγματικότητα η Πράσινη Συμφωνία, έχω αναλάβει να διασφαλίσω την έγκαιρη εφαρμογή του, της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει από 18 κράτη-μέλη το σχέδιο τους για την καθαρή ενέργεια. Τα υπόλοιπα εννέα μας έχουν ε, στείλει κάποιες ε, στρατηγικές, αλλά όχι ακόμα σχέδια. Γι' αυτό και θα στείλω επιστολές στους αρμόδιους υπουργούς, έτσι ώστε να τους ε, παροτρύνω να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Η πολιτική βούληση είναι πάρα πολύ σημαντική για να πετύχουμε τους στόχους μας, γι' αυτό και χρειάζεται η συνεισφορά όλων των κρατών μελών. Ε, αφού λάβουμε τα σχέδια θα τα αναλύσουμε έτσι ώστε να καταρτιστεί μία λεπτομερής ε, αξιολόγηση της κατάστασης μέχρι το φθινόπωρο του 2020. Εάν αυτό δεν επαρκεί, θα προτείνουμε πρόσθετα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, η συνεισφορά αυτή θα βοηθήσει τους φιλόδοξους στόχους ε, για την μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 50% και σχεδόν 55% μέχρι το 2030 και αυτό με υπευθυνότητα. Επίσης θα γίνει μια προσεκτική αξιολόγηση των ε, καλύτερων δυνατοτήτων ε, που έχουμε για να επιτύχουμε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο και γι' αυτό χρειάζεται να τεθούν στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την καθαρή ενέργεια. Θα κλείσω, αγαπητοί συναδελφοί, λέγοντας ε, δύο λόγια για την διεθνή διάσταση της, του σχεδίου αυτού. Ο ενεργειακός τομέας είναι ο σημαντικότερος και είναι εμβληματικός ε, για την προσπάθειά μας. Ε, αν δεν ε, καταφέρουμε να προσελκύσουμε τους σημαντικούς εταίρους σε αυτό και τους φορείς σε αυτό το θέμα, δεν θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στο Αμπουντάμπι, όπου συμμετείχα σε διάφορες διμερείς και Ανοιχτέ διασκέψεις και κατέστη σαφέ ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων. Η θέση της Ευρώπης που θα υιοθετήσουμε τους επόμενους μήνες θα καθορίσει την ε, παγκόσμια μετάβαση προς ε, την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εναρμονίσουμε την εξωτερική μας δράση με τις εσωτερικές μας κλιματικές φιλοδοξίες. Γι' αυτό στηρίζω τη δημιουργία της πράσινης ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία μας ε, με την περιοχή αυτή αλλά και με τους ε, γειτονές μας ε, στο Νότο και πρέπει να ενισχύσουμε και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να μεταδώσουμε τεχνογνωσία και να υιοθετήσουν και άλλοι τα ενεργειακά μας πρότυπα. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να σας έδωσα μια συνοπτική εικόνα των ε, πτυχών της Πράσινης Συμφωνίας και φυσικά με μεγάλη χαρά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ωστόσο να πω ότι βρισκόμαστε ακόμα στην ε, αρχή. της ε, προτάσεις θα πρέπει να ακολουθήσει σκληρή δουλειά, πολλές διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και με εσάς τόσο σήμερα όσο και τους ερχόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Thank you very much indeed for uh, your presentation. Σας ευχαριστούμε για αυτή την εισήγηση και για τις εξηγήσεις που δώσατε για το, η Πράσινη Συμφωνία και την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης ε, και που σταθήκατε και στην διεθνή διάσταση που είναι εξίσου σημαντική. Στρέφομαι στους συντονιστές. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, η κυρία Καρβάλιο. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και πάλι. για να παρουσιάσετε τα σχέδιά σας στην Επιτροπή Ήτρε για την Πράσινη Συμφωνία. Με χαρά βλέπουμε ότι η Πράσινη Συμφωνία έχει μια σφαιρική προσέγγιση, συμπεριλαμβάνει όλους τους κλάδους της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό όχι μόνο η ενέργεια, όχι μόνο η βιομηχανία να συμβάλλει στην Πράσινη Συμφωνία, όλοι οι κλάδοι να συνεισφέρουν. Έχω τέσσερα σημεία να θίξω. Πρώτον, ο κρίσιμος ρόλος της υλοποίησης των όσων έχετε ήδη στις υπηρεσίες σας Ήδη είχε εγκριθεί από την προηγούμενη επιτροπή το πακέτο οι με μέτρων για την καθαρή ενέργεια». Υπάρχουν πολλά μέτρα εκεί, πρέπει να ελοπιθούν από τα κράτη-μέλη. Τι σχέδια έχετε λοιπόν για την επιτάχυνση αυτής της εφαρμογής. Δεύτερον, το επίπεδο φιλοδοξίας σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Είναι σημαντικό για το ΕΛΚ να βασιστούμε σε μια εμπεριστατωμένη και λεπτομεριακή μελέτη αντικτύπου, αν μπορείτε να το σχολιάσετε και αυτό. Τρίτον, μιλήσατε για την έρευνα και την ανάπτυξη και πόσο σημαντικές είναι. Αλλά κυρίως αναφερθήκατε στις τεχνολογίες ε, που ήδη αναδύονται, υποδομές, υδρογόνο. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι αν θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας πρέπει να κινηθούμε και σε άλλες νέες τεχνολογίες. Δέσμευση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, για παράδειγμα, και άλλες τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στο πλαίσιο του πρόγραμμα Horizon Ευρώπη και ελπίζουμε να υπάρχει ο κατάλληλο ε, προπολογισμό για το ορίζον. Κάτι τελευταίο. Συνολικά για αυτή την ε, πράσινη μετάβαση χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, στο πλαίσιο ενός προπολογισμού που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς βλέπετε τη μετάβαση λοιπόν για την οικονομία και την κοινωνία μας, πώς θα εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις για αυτή τη μετάβαση στην οποία όλοι στοχεύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Νίκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Επίτροπε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και με ικανοποίηση βλέπω ότι σε αδρές γραμμές όλοι είπατε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε τα καλύτερα τα αποτελέσματα για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική. Κατά την προηγούμενη θητεία ε, υπήρχε μια πιο ήπια ε, παρουσία της Επιτροπής και θέλουμε να έχουμε πιο δραστήριο και ενεργό ρόλο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι σημαντικό αυτό που θέλουν οι καταναλωτές. Θέλουν να έχουν πρόσβαση ε, σε ένα απαραίτητο αγαθό που είναι η ενέργεια και σε προσιτές τιμές. Σε κάποιες περιοχές ε, της Ευρώπης ε, κάνει πολύ κρύο. Ο κόσμος θέλει να έχει πρόσβαση στην ενέργεια. Και μάλιστα σε φθηνή ενέργεια, προσιτή οικονομικά και θα ήθελα να ζητήσω να λάβετε υπόψη όλα αυτά που επιθυμούν οι καταναλωτές. Μετά πώς θέλετε να προσεγγίσετε αυτό το πρόβλημα που πλήττει πάνω από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, στην ενεργειακή ένδυα. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιμείνει πολλές φορές αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να υπάρξει τέτοια μνήα και στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά, οι νέες τεχνολογίες. Έχουμε τις νέες ε, ενεργειακές πηγές, ε, ανανεωσίμων, υδρογόνου και το καθεξής. Θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά ε, στο νομοθετικό μας πλαίσιο, αλλά κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο βάσει ενός ε, καταλόγου επιθυμιών και εμείς να ερχόμαστε εκ των υστέρων και φυσικά να βρισκόμαστε προεκπλήξεως γιατί δεν υπήρξαν διαβουλεύσεις ε, από πριν. Πρέπει να ξεχρονίσουμε τα δίκτυα φυσικού αερίου. Είπατε πρέπει να υπάρξει μετάβαση. Πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε χώρες όπου ε, σε χώρες όπου το φυσικό αέριο έχει πάνω από 30% του ενεργειακού μείγματος. Θέλουμε κι εμείς ε, να αντικαταστήσουμε και να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα. Η καλύτερη λύση θα ήταν ε, το ε, αέριο, είπατε. Υπάρχει το πρόβλημα της αποθήκευσης της ενέργειας που προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένω, δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή τη λύση από πλευρά ε, ε, ενεργειακή ασφάλεια. Τι θέση έχετε ω προ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναφέρει ότι κάποια έργα δεν μπορούν να υποφεληθούν χρηματοδότηση για το φυσικό αέριο. Πώ ε, θα λύσουν λοιπόν αυτέ οι χώρε το πρόβλημα τη απαλλαγή από τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαμπάγιοβα από την ομάδα Renew. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, αγαπητή Κάντρη, καλώ ήλθατε στην συνάντηση συνεδρίαση τη ομάδα Ήτρε για την παρουσίασή σα. Εμεί ε, είμαστε φυσικά υπέρ ενό φιλόδοξου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα. Θα δώσουμε μεγάλη λοιπόν έμφαση στο χαρτοφυλακιό σα ε, και άλλοι συνάδελφοι θα σας ε, θέσουν ερωτήματα γιατί είναι ειδικοί σε αυτό το ζήτημα. Επομένω από εμάς θα έχετε σίγουρα την αμέριστη στήριξή μας. Εν συντομία, ορισμένα ερωτήματα και οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν. Ε, μιλήσατε για τις κατευθύνσεις γραμμές για τα δίκτυα TNT. Σας ευχαριστούμε για αυτή την μνήα. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο έχει θέσει σημαντικές επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα χρηματοδοτήσουμε και θα διευκολύνουμε ενεργειακά προγράμματα που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς μας στόχους. Και χθε τα συζητήσαμε, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση το γεγονό ότι η Ολομέλεια υιοθέτησε τον Ιανουάριο θέση για τα TNT και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τι κατευθυντήριε γραμμέ ε, εγκαίρω για το PCIS είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε ε, ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλο ε, του χρόνου για την αναθεώρηση. Ε, θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετά νωρί, γιατί εμεί θέλουμε μια έγκαιρη πρόταση για αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών και θα πρέπει να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου ε, ο μηχανισμός του συνδέοντας στην Ευρώπη να βασίζεται σε εύρωστα ε, και ε, φιλικά προς το περιβάλλον κριτήρια. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν να επιταχύνετε τη διαδικασία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δεύτερον, ενεργική εξοικονόμηση στα κτίρια. Φυσικά έχουμε τεράστιες δυνατότητες εδώ. Στην τελευταία θητεία, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν ε, σε, ένα, μια αναθεωρημένη οδηγία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων που θέτει φιλόδοξους στόχους για την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης ε, των κτηρίων μας. Τι βήματα θα κάνετε ως Επίτροπος για να κινητοποιήσετε πλήρως ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις που χρειαζόμαστε σε αυτό το τομέα και πώς θα εντάξετε ευφυείς ψηφιακές λύσεις σε όλη αυτή την πρωτοβουλία τι νομοθετικές ή μη νομοθετικές ε, ε, προτάσεις μπορούμε να περιμένουμε από πλευρά σας. Μεταμιλήστε για τα ενεργειακά σχέδια ενέργειας και κλίματος. Σας ευχαριστώ και αυτό. Ένα ερώτημα μόνο. Πού εντοπίζετε τα κενά μεταξύ των σχεδίων αυτών και των στόχων που έχουμε θέσει. Και κάτι που είναι σημαντικό για τα κρατημέλη, πώς η Επιτροπή προσφέρει και παρέχει τεχνική συνδρομή για την αναθεώρηση ε, των σχεδίων. Επί του πρακτέου δηλαδή. Και κάτι τελευταίο, πώς συνεργάζεστε με άλλους ε, επιτρόπους για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικά σας θέματα. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να πείτε πολλά με τους επιτρόπους Τίμερμανς και Γκάμπριελ, αλλά και Μπρετόν και Βερστάγκερ. Τι μορφή λοιπόν παίρνει αυτή η συνεργασία και είστε τεθειμένοι να κάνετε περισσότερα για να συνεργαστείτε περισσότερο με άλλα χαρτοφυλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, θα κλείσουμε τώρα τον κατάλογο ομιλητών για το δεύτερο γύρο, γιατί ήδη έχουμε 20 συναδέλφου που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ελπίζω να είστε ήδη στον κατάλογο. Εντάξει, θα σας ε, βάλουμε. Κλείνει λοιπόν τώρα ο κατάλογος. Θα συνεχίσω με τον κύριο Νίμιστο, συντονιστή των Πρασίνων. Ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσίασή της. Η Πράσινη Συμφωνία είναι βασικό μέλημα της Κομισιόν και όλης της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή της, να δούμε τους στόχους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε βεβαίως είναι να δούμε τους στόχους του, μέχρι το 2030. Εκεί πιέζουμε πάρα πολύ για μία μείωση 55%. Ε, οι πράσινοι θέλαν παραπάνω, αλλά τέλος πάντων θέλουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου να μιλάει για 55%. Θέλουμε να μιλήσουμε επίσης για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή αποδοτικότητα και συγκεκριμένους στόχους. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε για τους νέους στόχους ως Κομισιόν και πώς θα κινηθείτε προκειμένου να υπάρξει εφαρμογή τους. Για να πετύχει η Πράσινη Συμφωνία ε, ως ε, βιομηχανική επανάσταση για να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει να δείξουμε και ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη για το κλίμα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει και νομοθεσία αλλά και χρηματοδότηση. Πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το πεδίο. Μιλήσατε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανακαίνιση κτηρίων. Ε, θα υπάρξει νομοθεσία για αυτά τα θέματα, πέρα από τη χρηματοδότηση βέβαια που χρειάζεται. Επίσης, μια και το δίκαιο για το κλίμα είναι βασικό θέμα για την Κομισιόν. Πώς από τα ενεργειακά θέματα θα αντιμετωπιστούν ε, στην νομοθεσία για το κλίμα, προκειμένου να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα. Αναθεωρείτε τους στόχους του 2030 και βάζετε και στόχους πριν το 2030, ούτω ώστε το δίκαιο για το κλίμα είναι πραγματικά, να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Εμείς οι πράσινοι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία. Πρέπει η Ευρώπη να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τώρα αμέσω. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ενδιάμεσες λύσεις, θα πρέπει από την απροθυμία και την, το, το δισταγμό να κινητοποιηθούμε και να εφαρμόσουμε νέους στόχους. Να τους θέσουμε και να τους εφαρμόσουμε. Αυτό είναι βασικό καθήκον της Κομισιόν και πρέπει να το κάνει τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάολο Μπόρκια από το ID. Καλημέρα, Επίτροπε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Το Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έφτασαν σε συμφωνία για τον καονισμό για την ταξονομία για την ποιοτική ταξινόμηση, όχι όμως δεσμευτική, της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων, ε, επενδύσεις που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και μη βιώσιμη. Και ο άνθρακας πήγε στις, ε, στον κατάλογο των επενδύσεων που δεν τις ε, προωθούμε. Μέχρι στιγμής η συμφωνία αυτή θα δίνει στην Κομισιόν τη δυνατότητα να καθορίζει τεχνικές παραμέτρους για να προωθήσει μια συγκεκριμένη ας πούμε οικονομική δραστηριότητα. Όχι να την απαγορεύσει, να την προωθήσει. Εσείς τι ρόλο βλέπετε ότι θα έχει το φυσικό αέριο στο μέλλον, δεδομένης της εισαγωγής που μας παρουσιάσετε σήμερα το πρωί. Το θέμα αυτού του φυσικού αερίου τέθηκε και από άλλο συντονιστή. Ποιες είναι οι προοπτικές σας για τη συμπερίληψη, πιθανή συμπερίληψη του φυσικού αερίου στην ταξινόμηση αυτή, τη φορολογική ταξινόμηση. Και τι θέση έχετε εσείς προσωπικά γι' αυτό. Ευχαριστώ. ECR. Ποσανόφσκι. Από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Χαίρομαι που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ενέργεια θα είναι ένα πολύ δύσκολο τεχνικό και οικονομικό θέμα. Έχει τεχνική και οικονομική διάσταση. Αν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικές ε, αλλαγές δηλαδή. Κατά την άποψή μου, μετά το 2030 οι περισσότερες χώρες θα έχουν κάποιο έλλειμμα. Λόγω της ε, σταδιακής ε, εξάλληψης ε, διαφόρων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής. Μέχρι στιγμής έχουμε μεγάλο δυναμικό. Δεν, δεν, μπορεί να περιμένετε, δεν μπορούμε να περιμένουμε βέβαια η, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αυξηθεί σημαντικά. Αλλά αν υπάρξει κινητικότητα μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κτλ, προφανώς και θα αυξηθεί η ζήτηση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε σχεδιάσει τίποτα για, αυτό το, για αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν σχεδιάζονται μία νυχτή. Χρειάζεται μακρόπνο σχεδιασμός. Μόνο και μόνο για να φτιάξουμε τις κατάλληλες υποδομές για την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτή είναι μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία. Αν θέλουμε να περάσουμε την ηλεκτροπαραγωγή που βασίζεται στον άνθρακα σε ηλεκτροπαραγωγή χωρί ε, άνθρακα. Χρειαζόμαστε σχέδια, πρέπει να φτιάξουμε τι υποδομέ, πρέπει να κάνουμε μελέτε αντικτύπου. Μετά το 2030 θα χάσουμε και πυρηνικέ εγκαταστάσει και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα. Για τα επόμενα 10 χρόνια μετά, τι σχέδια έχετε. Γιατί το 2030 είναι πρώτον θυρών, πρώτον πυλών. Η κυρία Κοντουρά από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για την κυρία Σίμψον. Ε, η μία είναι για την ενεργειακή φτώχεια ε, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ε, και τις δράσεις ε, για το κλίμα, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εκτιμήσουν στα ενοποιημένα εθνικά σχέδιά τους για την ενέργεια και το κλίμα, τα οποία έστειλαν μέχρι το τέλος του 2019, τον αριθμό των οικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια. Σας ρωτάω λοιπόν αν έχετε μία σαφή εικόνα για το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για το ποιες πολιτικές και μέτρα από αυτά που υιοθετούνται και εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της αξιολογούνται ως αποτελεσματικά. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχετε αποκομίσει από τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών. Επίσης, στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η Επιτροπή αναφέρει ότι κατά το τρέχον έτος θα παράσχει καθοδήγηση για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ενεργειακής παινίας. Στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λίγες ημέρες για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σας ζητάει συγκεκριμένα μέτρα και κατευθύνσεις και θα ήθελα να μας, να μας διευκρινίσετε ποιες πρωτοβουλίες ε, και συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να πάρετε. Το δεύτερο που αφορά τη δίκαιη μετάβαση στα νησιά, η μετάβαση αυτή σε καθαρή ενέργεια μπορεί όχι μόνο να συντελέσει σε μεγαλύτερη αυτάρκεια και ευημερία των νησιών, αλλά και να προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στις τοπικές ε, κοινότητές τους. Δεδομένων των αναθεωρημένων πολύ φιλόδοξων στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η εντολή της Γραμματείας θα λήξει τον Ιούνιο του 2020, προκύπτει η ανάγκη να δημιουργηθεί μια μόνιμη ευρωπαϊκή δομή ή όργανο για να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές απεξάρτησης από τον άνθρακα των νησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν σκοπεύει η Επιτροπή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να διασφαλίσει τη μελλοντική στήριξη της καθαρής και δίκαιας ενεργειακής μετάβασης στα νησιά και επίσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο της μετάβασης, θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να επικεντρωθείτε στην οικονομική πτυχή της ενεργειακής μετάβασης των νησιών, όπως είναι η γεωργία, η ηλία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι τοπικές βιομηχανίες, μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού μηχανισμού χρηματοδότησης έργων στα νησιά ή τη δημιουργία ενός ταμείου χρηματοδότησης ειδικά για τα νησιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο, τέλ, τέλος αυτού του γύρου σε έναν ακόμα συνάδελφο για ένα λεπτό γιατί πρέπει να φύγει για να πάρει το αεροπλάνο της. Εύα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτησή μου προς την Κομισιόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω επίτροπε που ήρθατε εδώ, ε, πολύ συγκεκριμένα τα όσα είπατε. Πώς ε, σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Φερρυπή, στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τους ίδιους στόχους για τις εκπομπές ε, σε αυτές τις χώρες, όπως προτείνει και για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι εγγύσεις θα έχουμε ότι θα τις σεβαστούν, χωρίς να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν στρεβλώσεις ε, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φτηνά ορυκτά καύσιμα που προέρχονται από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων των συντονιστών. Έχετε 10 λεπτά. Θα προσπαθήσω να, μέσα σε 10 λεπτά να καλύψω όλα τα θέματα. Η κυρία Καρβάλιο πολύ σωστά είπε ότι η Πράσινη Συμφωνία αφορά όλους τους τομείς. Αλλά στον τομέα της ενέργειας δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Έχουμε πολύ σημαντικές ε, συμφωνίες στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια και τμήμα της δουλειάς μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το πακέτο και όλα όσα έχουν συμφωνηθεί εφαρμόζονται. έχουμε και ένα πολύτιμο εργαλείο. Τα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος. Ο κύριος Στοσανόφσκι ρώτησε αν έχουμε κάποια εναλλακτική λύση, κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, κάποιο άλλο σχέδιο για να μας βοηθήσει να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Ναι, έχω δει σχέδια εθνικών προγραμμάτων από Είχαμε την προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2019 για να υποβάλουν αυτές τις, ε, αυτά τα σχέδια τα κράτη-μέλη και έχω δει λοιπόν κάποια σχέδια ήδη από κάποια κράτη-μέλη και εκεί υπάρχουν τέτοιες ιδέες. Για να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, της συμφωνίας, τα εθνικά σχέδια λοιπόν είναι το κλειδί. Είναι η νομοθετική βάση για την ε, συλλογική υλοποίηση των στόχων κλίματος και ενέργειας μέχρι το 2030. Τα εθνικά σχέδια θα μας επιβεβαιώσουν ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν διάφορες διαδικασίες. Καταρχάς υιοθετούν αυτά τα σχέδια και αντιμετωπίζουν το ερώτημα πώς θα αντικαταστήσουν τις πιο ρηπογόνες πηγές ενέργειας. Ούτως ώστε ώστε να πετύχουμε τους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε ποια κρατημέλη έχουν ήδη τέτοιες προτάσεις και μας έδωσαν τα σχέδιά τους. Είναι η Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, ε, Φιλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Κύπρος, Ουγγαρία και Τσεχική Δημοκρατία χθες. Είναι οι τρεις τελευταίες χώρες που μας υπέβαλαν τα σχέδιά τους. Εφτά κρατημέλη υποσχέθηκαν ότι θα μας στείλουν τα σχέδιά τους ε, μέσα στον Ιανουάριο επίσης από τα υπολοιπόμενα κρατημέλη. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε. για την υλοποίηση των στόχων του 2030. Μέχρι το καλοκαίρι του 2020 θα παρουσιάσουμε τα συνολικά σχέδια για, να, ε, για τη συνεισφορά το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των, στο, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ε, μέχρι το 2030, μείωση κατά 50% με στόχο να φτάσουμε το 55%. Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα, διάφορα μέσα, το ETS, την ενέργεια. Η ενέργεια θα εξασφαλίσει την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, μόνο από, μόνη της δηλαδή, η ενεργειακή αποδοτικότητα, κατά 45% και το υπόλοιπο το πετύχουμε τα υπόλοιπα μέσα, ETS κτλ. Έχουμε επίσης και νομοθεσία για τα δάση. Για τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή αποδοτικότητα θα αξιολογήσουμε τους της φιλοδοξίας των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. Έχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν αποκτήσει νέα κυβέρνηση και επομένως χρειάστηκε να παρατείνουν τις διαδικασίες. Μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα αξιολογήσουμε την επίπτωση της ενεργειακής νομοθεσίας και θα προτείνουμε αναθεώρηση των στόχων αν χρειάζεται. Έχετε ρωτήσει για τις πρωτοβουλίες ορισμένοι από εσά που δεν είναι άμεσα δική μου πρωτοβουλία, αλλά χρειάζεται να συνεργαστώ με συναδέλφους. Φαντάζομαι ότι εννοείται πρωτοβουλίες οι οποίες θα δημοσιευθούν ως Νούπο, τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου, όπως ε, το δίκαιο για το κλίμα, ε, βιομηχανική στρατηγική και σας επιβεβαιώνω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία στην ομάδα των δικών μου επιτρόπων υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Τίμερμαντς, αλλά και με τους υπόλοιπους επιτρόπους, αν υπάρχει θέμα που άπτεται της ενεργειακής πολιτικής ή της βιομηχανικής πολιτικής. Μαρτίνα, ανησυχείς ότι η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών των TEN ή των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας δεν είναι τόσο φιλόδοξη ε, όσο υποσχεθήκαμε. Θέλουμε να τηρήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Η Πράσινη Συμφωνία προβλέπει την αναθεώρηση των κατευθυντηριών γραμμών των TEN-E, δηλαδή των διευρωπαϊκών δικτύων ε, ε, ενέργειας, ως προτεραιότητα. Η αξιολόγηση έχει επιταχυνθεί και θα κάνουμε νομοθετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2020 για το θέμα αυτό. Ο στόχος είναι τα επόμενα, με τον επόμενο κανονισμό 10E να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 2050. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις έξυπνες ενεργειακές υποδομές. Το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει καινοτόμε τεχνολογίες και υποδοχή, έξυπνα δίκτυα, ε, πράσινα αέρια, ε, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, ε, αποθήκευση ενέργειας, και καινοτομία του κλάδου. Όλες αυτές οι μελλοντικέ λύσεις θα είναι στο τραπέζι μας. Ο κύριος Μπορκία με ρώτησε για την ταξινομία, ταξινόμηση της φορολογίας δηλαδή. Το συζητήσατε πολύ. Το συζητήσαμε το συζητήσατε γιατί είχατε και τριμερείς διαλόγους και τις ε, επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και οι οποίες είναι σημαντικές. Mm. Από μισό λεπτό. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το σύστημα ταξινόμησης για τις ε, πράσινες οικονομικές δραστηριότητες για να ε, δώσουμε κινήτρα για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες. Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται τμήμα της προσπάθειας που θα καταβάλουμε μέχρι το 2050. Αλλά βεβαίως ε, το ενεργειακό μείγμα το καθορίζει το κάθε κράτος μέλος. Ε, τι κάναμε λοιπόν για τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια. Ούτε τη συμπεριλάβουμε στον κατάλογο, δηλαδή ούτε την προωθούμε, δεν δίνουμε κίνητρα, αλλά ούτε την αποκλείουμε. Φυσικά, χάρη στα πυρηνική, στην πυρηνική ενέργεια, μειώνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Και πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι τμήμα του ενεργειακού του μείγματο για να πετύχουν του στόχου κλιματική ουδετερότητα. Όμως ε, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται πάντα η ασφάλεια, ιδιαίτερα στην ε, πυρηνική ενέργεια. Και όπως γνωρίζετε, τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν χρηματοδοτούν την κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων, όμως ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πυρηνική ασφάλεια, την διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και παρέχουμε στήριξη από εμπειρογνώμονες σε όλα τα κράτη-μέλη που το ζητούν. Επίσης, αναφερθήκατε μεταξύ άλλων στην ενεργειακή ένδυα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε στο Σώμα των Επιτρόπων διότι δεν θέλουμε να μείνει πίσω καμία περιοχή, καμία χώρα, καμία κοινωνική ομάδα. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο. Όμως ε, υπάρχουν παντού καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν μπορούν να πληρώσουν τους ε, λογαριασμούς τους, δεν μπορούν να πληρώσουν για θέρμανση, διότι συνήθως αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι πιο ακριβοί. Η ενέργεια κοστίζει. Και νομίζω λοιπόν ότι αν στηρίξουμε αυτό το κύμα ανακαινήσεων θα βοηθήσουμε όλους τους καταναλωτές να επωφεληθούν από αυτό και εκείνους που ζουν ε, σε κτίρια κοινωνικής στέγασης αλλά και τους πιο ευάλωτους. Όταν γίνουν ανακαινήσεις ε, στο κτηριακό απόθεμα όμως δεν υπάρχουν κονδύλια Υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί πολλή δουλειά από εμά και από τα κράτη-μέλη, αλλά κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους δημάρχους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν συνέργειες, καλές σχέσεις, ε, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς τι ποσοστό των ε, πολιτών σε κάθε χώρα δυσκολεύεται να πληρώσει τους ε, λογαριασμούς τους. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να λύσουν και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτό το ε, θέμα της ενεργειακής ένδυας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Όσοι έχουν ζητήσει το λόγο θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. 24 ε, παρεμβάσεις έχουν καταγραφεί. Σας παρακαλώ να μείνετε εντός ε, του ορίου του ενός λεπτού έτσι ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι και να έχει τη δυνατότητα η Επίτροπος να απαντήσει για άλλα 10 λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο γύρο, γύρο των ερωτήσεων με τον πρόεδρο Μπούζεκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε, που ήρθατε σήμερα. Είπατε ότι το 9% των παγκόσμιων εκπομπών προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πράσινη Συμφωνία. Και ταυτόχρονα είστε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 75% των ε, συνολικών εκπομπών της, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τον ενεργειακό τομέα, από τη βιομηχανία. Από τη βιομηχανία. Εμείς λοιπόν πρέπει να θέσουμε το καλό παράδειγμα, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να σωθεί ο πλανήτης. Το πρώτο στάδιο λοιπόν, δηλαδή η μείωση των εκπομπών, είναι το σημαντικότερο. Η μείωση μέχρι το 2030. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε φιλόδοξους στόχους, αλλά να φτάσουμε το 50% και όχι το 55%, διότι το 55% δεν θα αφήσει τους πολίτες ευχαριστημένους, θα οδηγήσει αυξήσει τιμών κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τερέζα Γκρίφιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. και σα ευχαριστώ πολύ που δεν είναι αυτή η τελευταία μου ευκαιρία να μιλήσω, διότι θα γίνει και άλλη συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα. Κυρία Σίμψον, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ε, η Μαρτίνα από το Renews είπε όσα ήθελα να πω, οπότε την ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε το 2015 τη συζήτηση για την ενεργειακή Ένδια και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω για το ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό μέσο, αλλά είναι μία μέθοδος προσαρμογής ε, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η νομοθεσία να είναι περιεκτική, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε διχασμό όπως έγινε χθε ε, στην ψηφοφορία. Γι' αυτό είναι πολύ απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση του σχεδίου και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα να μιλάτε για κοινωνική στέγαση και την ενεργειακή αποδοτικότητα που πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί εκεί. Επίσης υπάρχουν πολλοί ενοικιαστές ε, που δυσκολεύονται πάρα πολύ να ε, χρησιμοποιήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες για ανακαίνιση. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη θέρμανση των ε, σπιτιών τους. Εγώ προέρχομαι από το βορρά της ε, Αγγλίας, όμως ε, υπάρχουν χώρες του Νότου οι οποίες ε, υποφέρουν από την ζέστη το καλοκαίρι. Έχουμε και θανάτους από τον καύσωνα. Δεν πρέπει λοιπόν να διαχωρίζουμε μεταξύ θέρμανσης και ψήξης. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε όλε τι απαραίτητε πληροφορίε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υδρογόνο, υπάρχουν τρία είδη υδρογόνου. Το πράσινο, το μπλε ή το ε, γκρι. Δηλαδή, ε, το πολύ ε, οικολογικό, το μεσαίο και αυτό που βασίζεται σε άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει και ένας διαχωρισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ένα λεπτό λοιπόν σε ο καθένας σας και θα σας αποχαιρετήσουμε κυρία Γκρίφιν την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε σίγουροι. Περνάμε στον κύριο Γκιόρκ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω πως είναι προς το συμφέρον όλων να έχουμε ένα σχέδιο που θα στεφθεί με επιτυχία. Χρειάζεται όμως να γίνει βήμα-βήμα. Καταρχάς οι πολίτες πρέπει να έρθουν με το μέρος μας. Γι' αυτό χρειάζονται πλήρη ενημέρωση για όλες τις πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας, για το πώς η Πράσινη Συμφωνία θα επηρεάσει τις ζωές τους. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε μία λεπτομερή ανάλυση του πώς θα γίνει αυτή η ενημέρωση. Έπειτα, αυτή η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι προσιτή σε όλους. Και τρίτον, πρέπει να δούμε πώς ε, το κάθε κράτος μέλος θα αντιμετωπίσει τη μετάβαση αυτή. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, μεταξύ κρατών μελών. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στη Δυτική Ευρώπη ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ζει ε, σε ιδιωτικέ κατοικίε. Στην Ανατολική Ευρώπη τα πράγματα όμω είναι αλλιώ. Υπάρχουν άλλε δομέ και θα πρέπει να βοηθήσουμε με διαφορετικό τρόπο του πολίτε να ανακαινήσουν τα σπίτια του. Γι' αυτό κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι τα βήματα που θέλετε να ακολουθήσετε έτσι ώστε η Πράσινη Συμφωνία να χρηματοδοτηθεί ε, σωστά και να είναι οικονομικά προσιτή σε όλου. Ευχαριστώ πολύ. Η Πατρίσια Τόια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, Επίτροπε. Δύο παρατηρήσεις. Γιατί πρέπει να σας πω ότι είμαστε μεγάλος σας στη δουλειά σας εδώ η Επιτροπή μας. Επίσης, εάν δεν αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, δεν πρόκειται να, να υλοποιήσουμε τους ε, στόχους μέχρι το 2050 θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια, θα πρέπει να παρέμβει και να πάρει τον ηγετικό ρόλο, η Κομισιόν. Δεν μπορεί να περιμένει απλώς τα εθνικά σχέδια και να αφήσει τον μπαλάκι στη, στα κράτη. Είναι πολύ αδύναμη αυτή η πρακτική. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα, που είναι αδύναμα. Χρειάζεται ηγετικός ρόλος από πλευράς Κομισιόν. Αυτό ήταν το πρώτο. Και δεύτερον, αν θέλουμε να πετύχουμε ε, το 2050, πρέπει να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα τεχνολογικής φύσεως. Να λέμε, εντάξει, έχουμε τον ορίζοντα, ε, πρέπει να ανακαινήσουμε, ξέρω εγώ, τα κτίρια κτλ. Ε, αυτά είναι λίγα. Όλη η δραστηριότητα του ορίζοντα θα πρέπει να έχει σαν σκοπό την πρόθεση και τη διάδοση νέων τεχνολογιών. Γιατί χωρί αυτέ τι νέε τεχνολογίε δεν θα πετύχουμε του στόχου του 2050. Σα κάνω κριτικέ για να υλοποιήσουμε αυτού του φιλόδοξου στόχου και να μην το, του αφήσουμε γράμμα κενό περιεχομένου. Πρέπει να κάνει περισσότερα η Κομισιόν. Πολύ πιο αποφασιστικά να παίξει πολύ πιο έντονο ηγετικό ρόλο. Από το κύριε Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σε μια μεταβατική περίοδο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και εδώ, στην Ήτρε, σας ε, διαβεβαιώ ότι έχετε πολλούς φίλους και υποστηρικτές. για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις. Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω για την ε, υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας. Προτίθεστε να διασφαλίσετε μεγαλύτερο ε, επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των επιμέρους μηχανισμών που έχει τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των πράσινων στόχων και πιο συγκεκριμένα. Στο δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων εμπίπτει και το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κατευθύνουμε τον ορίζοντα προς την Πράσινη Συμφωνία. Μετά βέβαια έχουμε και το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προτίθεστε λοιπόν να βρείτε μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας ε, μεταξύ αυτών των χρηματοδοτικών μηχανισμών για να έχουμε και περισσότερες δυνατότητες προς ε, τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Λέει ο κύριος Καφ. Ε, σε ό,τι έχει να κάνει ε, με τα κτίρια. Η συνάδελφος Γκρίφιν έθεσε ένα αντίστοιχο ερώτημα. Σήμερα το πρωί εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα ξυπνήσουν ε, σε κρύα κτίρια γεμάτα υγρασία. Ζουν μέσα στην ενεργειακή ένδυα. Πρέπει να διαλέξουν άμεσα στην τροφή και στη θέρμανση. Για τα επόμενα χρόνια πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Έχουμε και την ε, οδηγία διατύπωση. Όμω, ε, εκεί στοχεύουν περισσότερο στα νέα κτίρια και στα δημόσια κτίρια. Πώς θα βελτιώσουμε ε, την κατάσταση στο απόθεμα κτηρίων και στα, στις ιδιωτικές κατοικίες ή ακόμα και στα δημόσια που συχνά παραμελούνται είναι βασικό κομμάτι τη ενεργειακή μετάβαση και εσεί θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει χρηματοδότηση. Ίσως μέσω συζητήσεων με διάφορους τομείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας δώσετε ακόμα μερικές λεπτομέρειες για τα σχέδιά σας. Τι θα κάνετε, θα έχετε νέους κανονισμούς για τα κτίρια ή θα στραφείτε περισσότερο στην αύξηση της χρηματοδότησης για να γίνει αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Σπυράκη. Thank Ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που είστε εδώ και πάλι μαζί μας. Πολύ σύντομα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον κατάλογο που έχει ήδη δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ορισμένα ποσά ε, για τα κάτι μέλη, για τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Δώστε μας ακόμα μερικές πληροφορίες. Ο μηχανισμός αυτός ε, θα είναι αναλογικός ή όποιος προλάβει. Και μετά θα θέλαμε οι περισσότερες ε, λεπτομέρειες για το πώς θα γεφυρώσετε το οικονομικό χάσμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στα προγράμματα για το φυσικό αέριο, το βιοαέριο και κουλουπού μετά το 2021. Ευχαριστούμε κύριο Κασνοντεύσκη. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα από μένα. Πρώτα λοιπόν για τα εθνικά σχέδια. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής είδαμε ότι τα σχέδια θα πρέπει να αντανακλούν τον νέο επίπεδο φιλοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμπλακεί περισσότερο στην εκπόνηση αυτών των σχεδίων στο μέτρο, στο μέλλον, συγγνώμη. Η Επιτροπή θα επηρεάσει πιο ενεργά τα κράτη-μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεύτερον, στον τύπο βλέπουμε ότι η Γερμανία δεν θα φτάσει, δεν θα πετύχει τον στόχο μείωση εκπομπών φέτος. Τον στόχο που είχε θέσει η Γερμανία το 2009. Σύμφωνα με περιβαλλοντικούς οργανισμούς, τώρα αυτό θα γίνει το 2030. Μάλλον μόνο η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ελλάδα θα πετύχουν τους στόχους του για το 2030. Τι θα γίνει τελικά αν δείτε ότι κανένα κράτος δεν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο τους. Αυτό βασίζεται στην ερώτηση του κυρίου Μπούζεκ. Εφόσον αυτή τη στιγμή ακόμα και μια τέτοια τεχνολογική δύναμη όπως η Γερμανία δεν είναι σε θέση να καλύψει το στόχο της. Και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι μόνο τρεις χώρες ε, θα τα καταφέρουν. Πόσο μάλλον να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο φιλοδοξίας. Τι θα γίνει αν τελικά δούμε ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζωρίνιο. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, που ήρθατε σήμερα εδώ. Όπως αναφέρθηκε, πρέπει να υλοποιήσουμε την Πράσινη Συμφωνία. και να είμαστε ηγέτιδα δύναμη στην απαλλαγή από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Χρειαζόμαστε εδώ την ενιαία αγορά πρέπει να λειτουργήσει καλά, δεν μπορούμε να έχουμε ενεργειακές νησίδες, ούτε να αφήσουμε χώρες ε, πίσω. Γι' αυτό πρέπει να ε, θίξουμε και το ζήτημα των διασυνδέσεων, που είναι κρίσιμη σημασία για να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. ήμουν ε, σκιώδης μαζί και με την ε, Τερίζα Γκρίφιν σε αυτό το φιλόδοξο ενεργειακό σχέδιο. Τι θα κάνετε εσείς για να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι διασυνδέσεις στο δίκτυο. Υπήρξε ένα ερώτημα για τη διασύνδεση του λιμένα του Σίνης στην Πορτογαλία με το δίκτυο φυσικού αερίου, βιοαερίου και ούτω καθεξής. Εσείς πώς θα αξιοποιήσετε το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης για να μπορούν και τα κρατημένη να είναι πιο φιλόδοξα στα εθνικά του σχέδια. Το Κοινοβούλιο, κατά τους τριμερείς ε, διαλόγους, ε, έθεσε σημαντικές απαιτήσεις. Τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν ε, στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων και ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συμβολή και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και στα εθνικά σχέδια δεν πρέπει να υπάρξει η ίδια προσέγγιση. Ευχαριστώ, κυρία Ένστ. Okay. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πίτροπε. Νομίζω πως συμφωνούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος χωρίς ε, μία αποδέσμευση από τη χρήση άνθρακα δεν είναι εφικτή, ούτε είναι λογική. Υπάρχουν ε, ορισμένες ε, περιοχές που βασίζονται στον άνθρακα, στην Πολωνία και αλλού. Και αν δούμε τι γίνεται με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, νομίζω πως θέλουμε να κάνουμε μαγικά για να τα καταφέρουμε. Έτσι να βρούμε το μαγικό φίλτρο για να γίνουν όλα καλά και όπως θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς θέλει θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτό το ταμείο όταν αρνούνται τα κράτη-μέλη να ε, συμμετάσχουν και αυτά. Επίσης, η χρήση του άνθρακα ε, στην Ευρώπη είναι μεγάλη. Για να αποδεσμευτούν οι επιχειρήσεις από τη χρήση άνθρακα θα χρειαστούν αποζημιώσεις σε τεράστια ποσά. Και σε άλλες χώρες ε, συμβαίνει το ίδιο. Στη Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλη χρήση άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τι θα κάνετε με τις αποζημιώσεις ε, για την αποδέσμευση από τον άνθρακα. Πού θα βρείτε τη χρηματοδότηση. Πώς αυτό είναι συμβατό με την ε, νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση έπειτα. Μια άλλη ερώτηση που έχω έχει να κάνει με την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. Το είπατε κι εσείς. Ε, η Τσεχία ήδη έχει ανακοινώσει ότι η πυρηνική ενέργεια θα συνεχίσει να προωθείται ως καθαρή ενέργεια. Πώς λοιπόν εσείς θέλετε να ε, πραγματοποιήσετε και την αποδέσμευση από άνθρακα και την από την χρήση πυρηνικής ενέργειας ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πίτροπε μπορώ και εγώ να συμφωνήσω με τα όσα είπε συναδελφός από του Σοσιαλιστέ. Η ενεργειακή ένδυα είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, αλλά και ε, αυτό θέλει την κατάλληλη χρηματοδότηση. Πώ μπορεί να γίνει. εμεί θέλουμε να γίνει πρώτα εκτίμηση αντικτύπου, έτσι ώστε αυτή η ανακοίνωση που προβλέπει 55% μείωση για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 να συνοδεύεται από εκτίμηση αντικτύπου, από λεπτομερή ανάλυση, έτσι ώστε να ξέρουμε τι κάνουμε. Έπειτα, το φυσικό αέριο. Θεωρώ πως το φυσικό αέριο το βλέπουμε κάπως αισιόδοξα. Τα... Η παραγωγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο μπορεί να ε, συνδυαστεί και με άλλα και με, την, ε, και με την χρήση υδρογόνου. Αν θέλουμε να γίνει σωστά ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό. Νομίζω όμω πω αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να συνδυαστεί, ε, να συνδυαστεί η αποδέσμευση από τον άνθρακα από την χρήση αυτή τη ενέργεια. Έπειτα θεωρώ πω στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλέ δυσκολίε στην κατάρτιση ενεργειακή πολιτική. Η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό κομμάτι τη εξωτερική μα πολιτική Πολλοί περιμένουν από μα και στην ε, Βόρεια Αφρική αλλά και σε άλλε περιοχέ να δημιουργήσουμε ε, συνεργασίε. και η ενεργειακή πολιτική θα πρέπει επίση να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι τη πολιτική γειτονία. γιατί η συνεργασία με τους γείτονές μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης, ε, κύριε Πίτροπε, ως Επίτροπος ε, Ενέργειας περιμένω να ε, χρησιμοποιήσετε ό,τι, όλη τη δύναμή σας και να είστε αυστηροί σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Ευχαριστώ κυρία Κομπουλανάτρη, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε Κάντρι για την ευρύτατη αυτή παρουσίαση. Ε, στην προηγούμενη θετία είχαμε στόχο 40%. Κάναμε πολλή δουλειά, αλλά τώρα έχουμε βάλει στόχο 50% και η πλειονότητα εδώ στο Κοινοβούλιο ήθελε 55%. Άρα πάλι πρέπει ε, να εργαστούμε πιο σκληρά και να έχουμε νέους, ε, νέα συνεργασία. Ιδάλλως δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ως θεσμικό όργανο. Εμείς εδώ θα σε στηρίξουμε. Για το 10E, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Εγώ διαπραγματεύτηκα τον μηχανισμό και το συνδέοντα στην Ευρώπη. Είναι πάντα δύσκολο να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, στην πράξη. Εάν πρώτα έχουμε τους στόχους, ε, μετά το, την οδηγια 10 TEN-E, μετά τη λίστα PCIS και μετά περνάμε στην υλοποίηση. Εμείς δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε κάτι το οποίο καταργείται ήδη σταδιακά, γιατί βλέπουμε καλύτερες τεχνολογίες διαβάζει ο κόσμος στις εφημερίδες και μετά νιώθει ανόητος εφόσον υπάρχουν καλύτερες τεχνολογίες και πιο οικονομικές γιατί εμείς να εμένουμε σε κάτι παροχημένο. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι η αγορά ήδη ξέρει καλύτερα. Βλέπουμε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να λάβει δράση. Αυτό μας επιτρέπει και να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες, αλλά ε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βούληση. Το ίδιο ισχύει και για τα κτίρια. Ήμουν σκιώδη ε, την προηγούμενη θητεία και ξέρω ότι πολλά πιστεύω μπορούν να μείνουν. Και η δίκαιη μετάβαση δεν έχει να κάνει μόνο με το ταμείο, είναι και πολιτική. Και για τα κτίρια δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτη ε, του οικήματο ή η οικογένεια που μένει. Μπορεί να είναι η πολυκατοικία, μπορεί να είναι η ευρύτερη γειτονιά που θα λύσει το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Πεκαρίνεν. Ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να μιλήσω φιλανδικά. Ευχαριστώ. Πριν από 10 χρόνια θέσαμε φιλόδοξους στόχους ε, στην Ευρώπη για το 2020. Θυμόμαστε το μείον 20, μείον 25%, συν 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στις μεταφορές συν 10% για τις ΑΠΕ. Αυτά για, για φέτος, έτσι, για το 2020. Επίσης, το 2018 είπαμε ότι τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε και το σύστημα εμπορίας εκπομπών, αλλά πλέον αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε αυξήσει τον ε, στόχο. Είμαστε πιο φιλόδοξοι. Πάμε στο μείον 50%. Πώς όμως καταμερίζεται, κατανέμεται αυτόν τον στόχο σε όλη την Ευρώπη. Και σε σχέση με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης ε, και τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές, θα θέσετε κοινούς στόχους για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί οι στόχοι θα κατανέμονται διαφορετικά ε, στις, ε, στα κράτη-μέλη όπως κάναμε στην αρχή, στο 2010, όταν αποφασίσαμε να κατανείμουμε τους εθνικούς στόχους για το 2020. Επιμερισμός λοιπόν του φόρτου σε σχέση με το ETS. Πώς θα γίνει όλο αυτό και αν θα θέσετε εθνικούς στόχους για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε, Χάν, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ξέρουμε ότι ε, η βιομηχανία ε, ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ε, ευθύνεται για την κατανάλωση του 30% της ενέργειας. Βιομηχανίες όπως η χαλιβουργία και η χημεία είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολη ε, κλάδη από περιβαλλοντική άποψη. Για να πετύχουμε το στόχο μέχρι το 2050 ή ακόμα καλύτερα μέχρι το 2040, οι εκπομπές ε, θα πρέπει φυσικά να περιοριστούν. Επειδή έχουμε και πολύ ε, μακροπρόθεσμους επενδυτικούς κύκλους, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε επενδύσεις σε παροχημένες λύσεις. Γι' αυτό και η ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει φυσικά να είναι πράσινη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα ποια μέτρα θα υιοθετήσετε συγκεκριμένα για να ενισχύσετε την απορρόφηση των ε, ε, τεχνολογιών RES και ETE e από ε, τη βιομηχανία και αν θα υπάρξουν νέα πρότυπα, νέοι κανόνες, νέα κίνητρα και μέτρα που θα επιβραβεύουν αυτούς που καταναλώνουν λιγότερο. Επειδή οι επιμέρου βιομηχανικοί κλάδοι έχουν ε, διαφορετικέ ανάγκε προκειμένου να κινηθούν προ την απομάκρυνση από τον άνθρακα, θα προτείνετε λύσει που θα μας επιτρέψουν να έχουμε γρήγορα μείωση των εκπομπών ε, χωρίς αυτό να επιφέρει ε, περί το κόστος. Μαρία Τζαν Μαρίνες. Μαρινέσκου, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Είπατε πολλά, τα οποία βεβαίως και στηρίζουμε. Όλα αυτά σας παρακαλώ να τα προασπίσετε και ενώπιον των συναδέλφων σας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ενεργειακό σκέλος θα τα αναλάβετε εσείς μιλήσατε για το φυσικό αέριο. Στο Ταμείο Δίκαιες Μετάβασης όμως δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, ε, παραγωγής, το κατανοώ, καύσης, εντάξει, αλλά για τη διανομή γιατί όχι. Η διανομή θα βοηθούσε ε, τη βιομηχανία, θα βοηθούσε την τηλεθέρμανση, θα βοηθούσε την θέρμανση κτηρίων. Μιλήσατε, μιλώντας για την ενεργειακή ένδυα μάλλον. Θα μπορούσατε να, να σχολιάσετε ακριβώς αυτό. Το Ταμείο δίκες Μετάβασης, Φυσικό Αέριο και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει χρήση του για τη διανομή. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Γκοντζάλης Κασάρης. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε Σίμψον, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, που είστε εδώ σήμερα μαζί μας και μας παρουσιάσατε τις προθέσεις σας για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει παρουσιαστεί, φυσικά και την υποστηρίζουμε και με προσήλωση θα εργαστούμε για την υλοποίησή της. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. η Ισπανία μέχρι το 2030 θα έχει ε, πετύχει όλους τους στόχους. Θα είμαστε καλός μαθητής. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα ε, η διασυνδεσιμότητα που ανέφερε ο κ. Ζωρίνιο. Είναι απολύτως απαραίτητο. Και χρειαζόμαστε επίσης ε, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να βρούμε τις απαραίτητες συνέργειες και να ενισχύσουμε όλους τους κλάδους. Σε αυτή τη στρατηγική λοιπόν μιλήσατε βεβαίως ε, για κάποια στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης είναι βεβαίως πράσινο, δεν είναι όμως αρκετά δίκαιο. Γιατί βρισκόμαστε εν μέσω μιας μετάβασης αλλά κάποιες χώρες δεν έχουν ε, ε, αναλάβει το μερίδιο της ευθύνη που τους αναλογεί. Όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν στη δίκαιη μετάβαση. Τέλος, αυτός ο κατάλογος PCI μπορεί να ελοποιηθεί χωρίς ε, να έχουν κάνει όλοι αυτό που πρέπει. Θα περιλαμβάνει και ε, τροποποιήσεις στην ομοθεσία. Ευχαριστώ, Σαν από τους πρασίνους. Μετά. Ευχαριστώ, Αν-Μαρή. Εγώ έπρεπε να ψηφίσω στην Envy, γι' αυτό είχε δώσει το δικό της όνομα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ και πάλι στο ρόλο των πολιτών. Ευχαριστούμε κυρία Σίμψον. Είπατε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η ε, Πράσινη Συμφωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Είναι μια ε, μάγνα κάρτα για τους ε, πολίτες. Έχει να κάνει και με την ενεργή κοινότητα και με τους ε, ενεργούς καταναλωτές που παράγουν ενέργεια και θα πρέπει ε, να δικαιούνται να εμπορεύονται για την ενέργεια που παράγουν στη γειτονιά τους από τον Bloomberg βλέπουμε που δεν είναι και τίποτα περιβαλλοντιστές και ε, ακτιβιστές είπαν ότι μάλλον μέχρι το 2027 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως από την ηλική ενέργεια, θα είναι πιο οικονομική από την λειτουργία, σε σχέση με τη λειτουργία των ε, ε, ε, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Τι μέτρα λοιπόν θα λάβετε εσείς για να διασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά θα υλοποιήσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Θα δώσετε κάποιες κατευθύνες γραμμές, ένα blueprint, θα κάνετε ε, συνέδρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούς από τη ΣΥΑΡ. Ευχαριστώ. Μέχρι τώρα, κανείς δεν μου έχει εξηγήσει πώς θα παράξουμε ε, αξιόπιστη ενέργεια και βιώσιμη οικονομικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με την ε, αιωλική και τα φωτοβολταϊκά. Ούτε το υδρογόνο είναι ενεργειακή πηγή, είναι ε, φορέας μεταφοράς ενέργειας. Το έχω πει πολλές φορές. Έχουμε ξεκινήσει χωρίς επιχειρηματική πρόταση. Χρειά... Μόνο τεράστια κονδύλια έχουμε. Εγώ πρώτο θα πω ότι θέλω την κατάργηση των νεκτοκαυσίμων, όχι όμω χωρί κάποια καλή εναλλακτική λύση. Επομένω, ξεκινήστε με μια ε, αξιολόγηση κινδύνου, των στομότερο δυνατόν. Πότε μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η κλιματική αλλαγή είναι η πρόκληση της γενιάς μας και χαίρομαι που ε, μπορούμε να εργαστούμε από κοινού σε αυτή την Επιτροπή προ όφελο των πολιτών και του πλανήτη. Δύο ερωτήσει. Μετά την παρέμβαση πολλών συναδέλφων που ανησυχούν όπως και εγώ ότι παρότι χρειαζόμαστε κάθε ευρώ που μπορούμε για την ε, δίκαιη μετάβαση αυτή τη στιγμή θα δώσουμε δεκάδες δις ευρώ για ε, έργα φυσικού αερίου που μάλλον είναι παροχημένα και θα μείνουν ε, και θα είναι άχρηστα στο μέλλον. Θέλω να σας καλέσω να κάνετε ό,τι μπορείτε για να υπάρχει έγκαιρη ανάληψη δράσης, να μην δαπανίσουμε χρήματα φορολογουμένων ε, για προγράμματα που δεν συνάδουν καθόλου με τους κλιματικούς μας στόχους. Μετά, και τα σχέδια της Επιτροπής και τα εθνικά σχέδια δράσης μιλούν για την ενεργική μετάβαση στις ανώνυμες πηγές ενέργειας, αλλά υπάρχουν χώρες όπου οι ΑΠΕ έχουν, δυσκολεύονται να απορροφηθούν στην αγορά. Όπως είδαμε, ας πούμε, στην Ουγγαρία, ότι ουσιαστικά έχουν απαγορεύσει την αιωλική ενέργεια και αυτό δεν επιτρέπει την ε, θέσπιση ευφυών δικτύων που θα βελτιώσει την κατάσταση για του καταναλωτέ. Μπορείτε λοιπόν να μα πείτε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, αξιολογήσει τα προσκόμματα στην, και τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά για συγκεκριμένε ΑΠΕ και πώ θα τα αντισταθμίσετε. Κύριο Χάιζελ, από τους Σοσιαλιστέ και Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σλοβακικά, μετρική μου γλώσσα. Επίτροπε, Άκουσα όλες τις ερωτήσεις και εσείς τις ακούσατε και μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει ένα χάσμα εδώ. Ε, τα κράτη-μέλη είναι διχασμένα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να εξοδεύουμε ευρωπαϊκά χρήματα για υποδομές φυσικού αερίου. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτοί, οι, αυτές οι υποδομές μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν για να χρησιμοποιηθούν, για να διανέμουν ε, καθαρό, μπλε ή πράσινο φυσικό αέριο. Εδώ ακούμε διαφορετικές πληροφορίες, ε, αντικρουόμενες που μας τις δίνουν οι λομπίστες. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας εξηγεί αν αυτές οι υποδομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα ε, και αν μπορούμε να, χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιηθούν τελικά ή μάλλον να γίνουν αυτές οι υποδομές ε, έργα τύπου PCI, δηλαδή ε, έργα κοινού ενδιαφέροντος για να χρηματοδοτηθούν για να χρηματοδοτηθούν σωστά. Γιατί ό,τι κάνουμε τώρα ε, το κάνουμε για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Η κυρία Νίμπλερ, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση που με απασχολεί τώρα τελευταία με όλη τη συζήτηση που έχει γίνει για τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Εσείς ως επίτροπο, ε, πώς μπορείτε να ασκήσετε επιρροή έτσι ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να παραμείνει οικονομικά προσιτή. Ε, το σχέδιο του Green Deal θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η ενεργειακή μετάβαση ε, προϋποθέτει και φτηνό ρεύμα ή οικονομικό προσιτό ρεύμα. Γι' αυτό λοιπόν έχω μια παράκληση εσείς και οι συνάδελφοί σας να ε, διεξάγετε μία, εκτέλεση, μία εκτίμηση αντικτύπου έτσι ώστε κάθε μέτρο που θα συνοδεύσει την Πράσινη Συμφωνία να μην είναι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον αλλά να συνυπολογίζει και τις ε, επιπτώσεις στην αγορά, στους πολίτες και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα, Επίτροπε. Σας ευχηστώ την προσοχή σε δύο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να τεθούν εάν η Κομισιόν θέλει να μιλήσει σοβαρά για την Πράσινη Συμφωνία. Ο ρόλος και οι προθέσεις της ε, ενεργειακής βιομηχανίας. Πριν ε, δύο εβδομάδες μια γερμανική εταιρεία ε, θα κάνει σοβαρές επενδύσεις στην Αυστραλία Αυτό θα τα ακούμε ε, όλο και περισσότερο τους επόμενους μήνες. Για μια καλή πράσινη συμφωνία θέλουμε λιγότερες τέτοιου τύπου συμβατικές υποχρεώσεις και θα πρέπει να προωθήσουμε ε, εταιρείες που πραγματικά επενδύουν στην πράσινη ενέργεια. Τι άποψη έχετε. Σε μια, με βάση μια ε, σοβαρή έκθεση οι ισχύουσα, ισχύουσες υποδομές φυσικού αερίου είναι ικανές ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικέ ε, ανάγκες φυσικού αερίου στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθε όμως ε, μόνο 17 από 72 ε, ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της ιδέας. Γιατί δεν θέλετε να έχετε κριτήρια PCI Πού είναι η φιλοδοξία σας, χρειαζόμαστε περισσότερη φιλοδοξία για να πετύχουμε μια πραγματική ενεργειακή επανάσταση. Οι τρεις τελευταίες ε, παρεμβάσεις, ο κύριος Μπλός από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Έχουμε μελέτες αντικτύπου. Προβλέπονται. Για να αξιολογήσουμε κυρίως τι είδους στόχους χρειαζόμαστε για το 2030. Αυτές οι μελέτες αντικτύπου βασίζονται στα εθνικά σχέδια ενέργειας και κλίματος. Έχουμε πολλές χώρες που δεν έχουν ακόμα υποβάλει όμως τα εθνικά του σχέδια. Αυτό επηρεάζει το χρονοδιάγραμμά σας για τις μελέτες αντικτύπου και επηρεάζει το χρονοδιάγραμμά σα για να θέσετε τους στόχους για το 2030. Δεύτερη ερώτηση για το υδρογόνο. Μιλάμε πολύ για το υδρογόνο. Ε, υπάρχει ζήτηση για υδρογόνο από πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ξέρουμε όμω ότι για να έχουμε πράσινο υδρογόνο, ε, αυτό είναι πολύ ενεργοβόρο και το δυναμικό που χρειάζεται για τέτοια ποσά υδρογόνου ε, το δυναμικό δεν υπάρχει ακόμα. Επίσης υπάρχει και θέμα μεταφοράς. Έχετε προβολές για, το, για τις ανάγκες σε πράσινο υδρογόνο και επιπλέον από πού θα προέλθει. Πού θα βρούμε δηλαδή αυτό το υδρογόνο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος μας μιλάει πάντα για την ε, κλιματική κρίση, η οποία θα μας ε, πλήξει σαν ένα κύμα σε 20-30 χρόνια και πρέπει να την προλάβουμε, να την ανασχέσουμε. Μέχρι το 2030 η μείωση του 50-55% είναι αρκετή για να αντικρούσουμε αυτό το κύμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει κυρία Λίτση. Εγώ εξελέγην πριν από λίγους μήνες. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, γιατί το θέμα της ενέργειας είναι οριζόντιο και αφορά πολλούς άλλους φακέλους που εξετάζει η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Ήτρε, ε, το Horizon, τον Ορίζοντα και πολλά άλλα. Και η κοινωνία των πολιτών ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα της ε, ενέργειας εν γέννη. Κατάλαβα ότι εδώ στην αίθουσα αυτή πολλοί συνάδελφοι θέλουν να γίνει μια μελέτη αντικτύπου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε ως συνομοθέτες σε πολλούς τομείς θα πρέπει να βασίζονται κάπου, σε ένα έγγραφο που θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Γιατί ε, μιλάμε για μεγάλα ποσά τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι. Πέρα από αυτά τα γενικά σχόλια, του γενικού προβληματισμού, ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο του Green Deal, τη Πράσινη Συμφωνία και όλων όσων ακούστηκαν σύστημα, ε, σήμερα, ποιο είναι ο ρόλο που θα δώσει η Κομισιόν στις ενεργειακές κοινότητες. Γιατί υπάρχουν διάφορα κινήματα ε, σε διάφορες ε, περιοχές και σε διάφορα κράτη που δεν έχουν λάβει ακόμα αυτή την οδηγία. Ποια θα είναι η σχέση σας, η αλληλεπίδρασή σας με αυτές τις ενεργειακές κοινότητες. Και οικονομικά και τεχνικά, ας πούμε, τι δράσεις μπορείτε να προωθήσετε ε, όταν ε, μιλάμε για φορείς ιδιωτικούς, όπως αυτές οι ενεργειακές κοινότητες. Η κυρία Τουσάν. Θα ξαναθέσω ένα ερώτημα που έχω ξαναθέσει. Γρήγορα θα έχουμε νομοθεσία. Χαιρόμαστε γι' αυτό, για τα θέματα που συζητάμε. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Υπάρχει διαφάνεια στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις για αυτόν τον κατάλογο των PCI των έργων κοινού ενδιαφέροντος. ενδιαφέροντος. Ξέρω ότι ξεκινήσατε τις συζητήσεις ε, και θα συζητήσετε το πέμπτο έργο του καταλόγου. Μου το επιβεβαιώνετε ότι θα αρχίσετε τις συζητήσεις γι' αυτό. Πότε θα μας ενημερώσετε εμάς για τις εξελίξεις ε, των συζητήσεων για αυτόν τον κατάλογο και για τα έργα τα οποία θα μπορούσαν να πιθανώς προβληματικά. Και τρίτο ερώτημα, πάντα για τη διαφάνεια, είναι το θέμα των κριτηρίων. Θα βασιστείτε σε ποια κριτήρια ακριβώς για να γίνουν αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Τουσά. Ε, ο κύριος Φούξλαντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Βλέπω την, το πάθος τη δέσμευσή σας ε, για την πράσινη ατζέντα. Το ΕΛΚ σας ενθαρρύνει να προωθήσει το 50%, όχι το 55%, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς οι σοσιαλιστές διαφωνούμε. Νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο 55%, γιατί νομίζουμε ότι αυτό χρειαζόμαστε, τουλάχιστον για να σεβαστούμε τη Συμφωνία του Παρισιού, την οποία υπογράψαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστηρίζει και τα κράτη-μέλη την υπέγραψαν. Το 50% δεν συμφωνεί με, το, με τη Συμφωνία του Παρισιού. Είμαστε αντίθετοι. Μαζί με την ε, πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπέρ του 55%. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα λοιπόν. Και θέλω να το, βάλουμε, να το λάβουμε και αυτό υπόψη τη συζήτηση. Δεύτερον, για το κανονισμό 10E των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργεια. Το αναθεωρήσατε. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά ανησυχώ για το εξή κάποια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Μόλις υιοθετήσουμε τον κατάλογο των PCI. Ε, μιλάμε για ε, project ε, φυσικού αερίου ύψους 29 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα πρέπει όμως να κλειδωθούμε και να δεσμευτούμε σε έργα που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα και προωθούν τα ορυκτά καύσιμα για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Θα πρέπει για να επηρεάσουμε τον κατάλογο των PCI και να ε, υποστηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αναθεωρήσουμε προηγουμένως τον κανονισμό ταινί. Πώς πρόκειται να προχωρήσετε σε σχέση με αυτό το θέμα. Τελευταία ε, παρέμβαση από το Ρινιού. Ο κύριος Γκροσέλ. Είμαι υπέρ των ε, στόχων των νεώσιμων πηγών ενέργειας η ενέργεια επηρεάζει όλες τις πτυχέ της μοντέρνα ζωής. Γι' αυτό περιμένω από την Κομισιόν ε, αξιόπιστα και ολιστικά σχέδια για να υλοποιηθούν οι στόχοι. Ε, όταν υπάρχει ένα μικρό λάθος, ε, το σύστημα παροχής ενέργειας μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις και τεράστια επιπτώσεις στην οικονομία. Θα υπάρχει συγχρονισμός, θα υπάρχει εναρμονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και κυρίως με, και με τις χώρες της ε, γειτονίας μας. Γιατί στο ενεργειακό σύστημα, ξέρετε ότι στην ενέργεια μάλλον, οτιδήποτε συμβαίνει στους γειτονές μας μας επηρεάζει άμεσα. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε. Πέρα από τους στόχους 50 ή 55, χρειαζόμαστε ε, ισχυρά, αξιόπιστα σχέδια για το πώς θα το πετύχουμε αυτό το 50%. Και έπειτα δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα λάθος στο, ε, στο κύκλωμα ανεφοδιασμού σε ενέργεια παροχής ενέργειας. Ήσασταν τελευταίος, αλλά σημαντικός βεβαίως. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος, πολλά από τα θέματα την οριζόντια. Σε ορισμένε παρεμβάσει, μιλάτε για τους κλιματικούς στόχους, για την ενεργειακή μετάβαση, για τον κατάλογο PCI είχαμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά και το Δεκέμβριο μαζί σα και αποφασίσαμε μαζί ότι το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία. Υπάρχουν όμω και πολλέ ε, ε, συγκεκριμένε ερωτήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 15 λεπτά, γιατί έχουμε χρόνο. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα πρέπει και άλλες ερωτήσεις, θα πρέπει να επανέλθετε. Αν έχετε και οποιασδήποτε άλλες δικές σας παρατηρήσεις, βεβαίως να τις ακούσουμε. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Εδώ είναι μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό αυτό. Ξέρουμε ότι όλοι προερχόμαστε από διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε ε, και από διαφορετικά κράτη-μέλη και άρα είναι θεμητό να έχουμε διαφορετικέ απόψει. Και η ενεργειακή πολιτική είναι μία από τι πολιτικέ που ενδιαφέρει απίστευτα του πολίτε. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το κλίμα και το περιβάλλον μέσω τη ενέργεια. Είναι θέμα λοιπόν ευθύνη και πρέπει να. Ακριβώ επειδή υπάρχει ευθύνη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτού του πολύτιμου πόρου και ότι έχουμε προσιτέ τιμέ και για του καταναλωτέ και για τι επιχειρήσει. Ο κύριος Μπούζεκ ξεκίνησε αυτό το γύρο. Με ερωτήσει για το αν είμαι σίγουρη ότι η αύξηση του στόχου για, τους, δηλαδή για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, αν αυξήσουμε τη φιλοδοξία, αν πάμε λέει, στο 50% ή στο 55% ας πούμε ακόμα περισσότερο, θα τα καταφέρουμε. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο αφετηρίας. Αν κάνουμε ό,τι συμφωνήσαμε σε επίπεδο ενέργειας, χάρη και μόνο στην ενέργεια, θα έχουμε μείωση των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 45%. Ορισμένοι με ρωτήσατε αν περιμένουμε ακόμα τα εθνικά σχέδια κλίματος και ενέργειας. Και στο μεταξύ δεν κάνουμε τίποτα. Ποια είναι η εξήγηση για το ότι δεν υπάρχουν ακόμα τα τελικά σχέδια από όλα τα κράτη-μέλη. Είναι ότι υπήρξαν σοβαρές διαπραγματεύσεις αφού οι κυβερνήσεις πρότειναν τα προσχέδια αυτών των σχεδίων, των εθνικών σχεδίων. Και πολλά κράτη-μέλη μετά από αυτές τις διαπραγματεύσεις αποφάσισαν να αυξήσουν τους, φιλοδοξίε τις φιλοδοξίες και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί υπάρχουν εθνικές διαδικασίες οι οποίες κρατάνε κάποιο χρόνο. Έτσι. Ε, για να πάρετε όμως, για να αυξήσετε τους στόχους πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται χρόνος. Και πρέπει να υιοθετηθεί τελικά επίσημα το τελικό κείμενο είτε από την κυβέρνηση είτε από το κοινοβούλιο σα. στο κοινοβούλιο τη χώρα δηλαδή. Θα πρέπει τα σχέδια να είναι ξεκάθαρα. Επίσης με ρωτήσατε αν εξαλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα. Ε, το λιγνίτι, την τύρφη, α, το λιθάνθρακα, ε, όλα τα ορυκτά καύσιμα. Πώς θα πετύχουμε το να έχουμε, ας πούμε, επαρκή ενέργεια. Κοιτάξτε, εμεί στον τομέα τη ενέργεια έχουμε φιλόδοξου στόχου. Θα πρέπει και οι υπόλοιποι τομεί να κάνουν αυτό που του απόκειται. Έχουμε το πακέτο καθαρής ενέργειας και υπάρχει μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να υπάρχει συνδυασμός των διαφορών τομέων. Μεταφορές, ε, στον τομέα της θέρμανσης και της ψήξης, να λαμβάνουμε υπόψη μας συνολικά σε ένα συνολικό πλαίσιο όλα, όλους τους τομείς. Και να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφορες ε, βιομηχανίες. Εκεί που δεν μπορούν ή δεν αρκεί, ας πούμε, η ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης, εδώ ακριβώς μπαίνει το θέμα του υδρογόνου που έχει τεράστιο δυναμικό ε, στην ε, μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Το ανανεώσιμο υδρογόνο μπορεί να στηρίξει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης έχει τεράστιες δυνατότητες ε, ενεργειακής αποθήκευσης. Μας βοηθάει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στις μεταφορές. Στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Ε, γιατί μιλάμε εδώ για, μια, για ένα κλάδο που έχει πάρα πολλές εκπομπές, έτσι, μεταφορές. θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι φιλοδοξίες μας είναι ψηλότερε από τις σημερινέ. Χάρη σε όλες αυτές τις συνδυασμένες προσπάθειες. Συνάντησα πολλούς από εσά στο παρελθόν και εσείς με ρωτήσατε για τις ε, διασυνδέσεις. Και συμφωνώ ότι ο ρόλος των ε, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικός. Μας βοηθάει να εντάξουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και δημιουργεί ε, μεγαλύτερες περιφερειακές αγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό όλες οι συμφωνίες οι οποίες έχουν ήδη συναυτεί να εφαρμοστούν. Επίσης θα υπάρχει δυναμικό των ε, σημείων διασύνδεσης για τις ε, διασυνοριακές περιοχές. Τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν είναι έτοιμα να, ακόμα, θα πρέπει να λάβουν δράση. Θα πρέπει να είναι έτοιμα σε πέντε χρόνια. Θα πρέπει να εφαρμοστούν λοιπόν σωστά αυτά τα σχέδια δράση, ούτω κάθε χρόνο η, να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο το δυναμικό των διασύνδετών, των interconnectors. Επίση, θα πρέπει να περιοριστούν οι επιδοτήσει στα εργοστάσια εκτοπαραγωγή που χρησιμοποιούν ακόμα τον άνθρακα και να περιοριστούν στο ελάχιστο, στο αναγκαίο. Ορισμένοι ε, είπατε ότι μερικέ φορέ είναι εύκολο να αντικαταστήσουμε τον άνθρακα με το φυσικό αέριο σε ορισμένου τομεί. Ε, και θα μπορούσε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση αυτή. Έχουμε και άλλα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία βοηθούν ε, ε, την ανανέωση των υποδομών τηλεθέρμανσης, του district heating. Υπάρχουν κάποιοι κανόνε, υπάρχουν και εξαιρέσεις όμω για ορισμένα κράτη-μέλη για, το, για την τηλεθέρμανση, το district heating. Για τη χρηματοδότηση των έργων φυσικού αερίου και το ρόλο του φυσικού αερίου κατά την μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση. Ο τέταρτος κατάλογος με έργα κοινού ενδιαφέροντος υποβλήθηκε από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για να υλοποιήσουμε τους στόχους μέχρι το 2050 και για να γίνει αυτό θα πρέπει ε, να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του φυσικού αερίου. Ε, ο πιο δύσκολος τομέας σε αυτή την ε, περίπτωση είναι ο τομέας ε, των μεταφορών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και τον πέμπτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. Ε, και το Δεκέμβριο είχαμε ακούσει, είχαμε δεσμευτεί μάλλον, να εμπλέξουμε περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εμπλέξουμε τις ε, πιο αρμόδιες ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπές στις συζητήσεις αυτές για, τους, ε, για τις ανάγκες υποδομών σε ποιες ευρωπαϊκές περιφέρειες και στην αξιολόγηση των έργων αυτών και την αντιπαραβολή τους με τις ανάγκες. Επίσης, ο κανονισμός TEN-E συνδέεται με αυτό. Ο πέμπτος κατάλογος έχει ξεκινήσει και στην, στα, για τα υπόλοιπα που δεν, project που δεν τα έχουμε συζητήσει, θα κάνουμε μελέτες. Μέχρι τα μέσα του 2020 θα τις έχουμε έτοιμες. Και θα ενσωματώσουμε όλα τα project που δεν έχουμε ακόμα συζητήσει και αποφασίσει για αυτά στον κατάλογο. Επίσης, πολύ με ρωτήσατε τι γίνεται με το δίκτυο ε, ενέργειας. Ε, μου είπατε ότι σε διάφορα νοικοκυριά έχουμε διαφορετικές λύσεις ενεργειακές. Παραδείγματο χάρη και διαφορετικές ανάγκες. Παραδείγματο χάρη ε, τα νοικιασμένα σπίτια έχουν άλλες δυνατότητες ή άλλες ανάγκες από τα ιδιόκτητα. Και κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του νομικό πλαίσιο, μπορεί να βοηθήσει τις κοινότητες, καταρχάς ε, για το ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθώντας τον επιμερισμό των καλών πρακτικών. Το κύμα ανακαινήσεων που έχει προαναγγελθεί στον τομέα των κατοικιών, γιατί το 40% των ενεργειακών αναγκών ε, καταναλώνεται για την ε, θέρμαση και ψήξη των κατοικιών. Θέλουμε καταρχάς ε, επιπλέον χρηματοδότηση για την ανακαίνιση. Τα ευνοϊκά χαμηλότοκα δάνεια δεν αρκούν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε ποια είναι όλα τα φράγματα που εμποδίζουν την ανακαίνιση των κτηρίων. Θα δούμε λοιπόν ε, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι τοπικέ αρχέ θα πρέπει να συνεργαστούν, ούτω ώστε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα ε, για να αυξηθεί το κύμα αυτό ανακαινήσεων και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανακαίνωση τομέων ειδική προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, όπω είναι τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Γιατί όταν εξοικονομήσουμε ενέργεια σε αυτό το επίπεδο, αυτό θα είναι πολύ επωφελές για τη δημόσια υγεία, αλλά και για την κοινωνική στέγη. Και για τα νοικιασμένα σπίτια θα βοηθήσουμε τις ανακαινήσεις αν μοιραστούμε τις καλές ε, πρακτικές. Παραδείγματος χάρη, έχουμε σπίτια στην Ανατολική Ευρώπη που χτίστηκαν δεκαετή του 80. Αν τα ανακαινήσουμε αυτά τα σπίτια, θα καταναλώνουν 40% λιγότερη ενέργεια από ότι τα μη ανακαινισμένα ίδια. Και βεβαίως θα μειωθεί και ο λογαριασμός ε, των ΔΕΚΟ, της ΔΕΗ. Μια ερώτηση για την ε, δίκαιη μετάβαση και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ότι δεν έχουμε το μαγικό ραβδάκι που θα λύσει το... όλα μας τα προβλήματα. Χρειάζεται να βοηθήσουμε κι άλλο τις περιφέρειες εκείνες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στο να ξεκινήσουν. Αυτές οι περιφέρειες ε, που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα. Και γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν κάθε μεγάλη μετάβαση σήμαινε πως ε, θα έμεναν αναγκαστικά πίσω ορισμένες ε, περιοχές. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η Πράσινη Συμφωνία να πετύχει να πιάσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τις ε, περιοχές αυτές να βρουν θέσεις απασχόλησης, να βρουν νέες λύσεις. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κρατημέλη, κυβερνήσεις θέλουν βοήθεια έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουν δράσεις που θα αποτρέψουν την απώλεια θέσεων απασχόλησης στις ε, περιφέρειες αυτές. διότι η πράσινη ενέργεια δημιουργεί μεν θέσεις απασχόλησης, αλλά από περιοχή σε περιοχή οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές. Επίσης, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να βοηθήσουμε την ε, κατάρτιση των εργαζομένων, να λάβουμε διάφορα μέτρα ανακατανομής του εργατικού δυναμικού. Και σίγουρα τα 7 πρώτα χρόνια θα είναι το αρχικό στάδιο. Ο στόχος μας είναι ε, στο 2050, το οποίο είναι αρκετά μακριά. Το 2050 απέχει το ίδιο με το 1990, οπότε μπορείτε να δείτε τη σχέση μεταξύ ε, του χρόνου που χρειάζεται. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε λογικά μέτρα, λογικές λύσεις για τη μετάβαση αυτή. Θα ήθελα τώρα να επιστρέψω στους φιλόδοξους στόχους μας. Ε, και πρέπει να επαναλάβω ότι ό,τι κάνουμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη, για τις κυβερνήσεις. Θέλουμε να ηγηθούμε, να δώσουμε το καλό παράδειγμα και στον υπόλοιπο κόσμο όμως. Γι' αυτό και ο ενεργειακός διάλογος με τους βασικούς εταίρους μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Θα ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος με τις Ηνωμένε Πολιτείες φέτος. και με την Κίνα και με την Αφρικανική Ένωση. Και ρωτήθηκα τι θα κάνω με τα κράτη των Βαλκανίων. Θέλω να απαντήσω ότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και τις γειτονικέ μας χώρες να αποδεσμευτούν από τον άνθρακα στην βιομηχανία τους. Η Προεδρία της Κροατίας έχει μάλιστα θέση ως προτεραιότητα την ε, πρωτοβουλία για τα πράσινα νησιά και την ε, πρωτοβουλία για τα Βαλκάνια. Οπότε λοιπόν ε, θα συνεργαστούμε στενά με την Προεδρία για τους στόχους αυτούς. Και Επίση, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε όσο το δυνατόν ε, περισσότερους ομοειδεάτε για να συνεργαστούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, συνάντηση. Με τα χαρά να απαντήσω και διμερώς στις ερωτήσεις Σα uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτροπα, για τις απαντήσεις σας. Φυσικά και θα είμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία μαζί σας, είτε και διμερώς, είτε και μέσω διαφορών εκδηλώσεων. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε τρία λεπτά θα ξεκινήσει η ακρόασή μας για τον ορίζοντα Ευρώπη. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε Κάντε λίγη υπομονή. Οι υπόλοιποι παρακαλείστε να αποχωρήσετε ήσυχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και τη συμμετοχή σας, την ενέργο συμμετοχή σας. Dear colleagues, uh, if you are ready, I would propose to start. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε την ακρόαση, διότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις να ακούσουμε. Θα ακολουθήσουν αρκετές παρεμβάσεις και όλας, διότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό για εμάς και την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω θερμότατα τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε έξι προσκεκλημένους σήμερα και θα ήθελα λοιπόν εκ μέρους της Επιτροπής Ήτρε να σας καλωσορίσω και να καλωσορίσω και το κοινό που μας παρακολουθεί σήμερα και τους συνάδελφους της Ήτρε που βρίσκονται εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σημερινή συνεδρίαση με μια δημόσια κρόαση για το στρατηγικό σχεδιασμό του ορίζοντας Ευρώπη αποστολές και εταιρικέ σχέσεις. Θα εστιάσουμε σε αυτό στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για το πρώτο στρατηγικό σχέδιο του επόμενου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία. Τον ορίζοντα Ευρώπη δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία ισχυρή και φιλόδοξη θέση για το πρόγραμμα αυτό, δεδομένου ότι η έρευνα και η καινοτομία θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, για τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Επίσης, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας μας για την Πράσινη Συμφωνία, αλλά και για άλλους πολύ σημαντικούς στόχους της Ένωσης, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση, οι καλύτερες ε, τεχνολογίες στην Ένωση και άλλα, ζητάμε έναν επαρκή προϋπολογισμό και η επίσημη πρότασή μας ήταν 120 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα, δηλαδή 8% παραπάνω από την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή μας ατελάσσει πολύ συχνά απόψεις και σε επικοινωνία με την Κομισιόν για, τον, τη στρατηγική εφαρμογή του προγράμματος. Έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το θέμα των εταιρικών σχέσεων και των ε, αποστολών μας και για τους πρώτους μήνες του 2020 θεωρούμε πως ε, έχει μεγάλη σημασία το τι θα γίνει. Θα καθορίσουν το μέλλον. Ο ορίζοντας Ευρώπη δεν ε, υπήρχε στο, στα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο. Οι αποστολές του ορίζοντα Ευρώπη, μάλλον. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ενσωματωθούν και είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες, είναι μεγάλο το πεδίο εφαρμογής. Θα ακούσουμε λοιπόν για δύο από αυτές τις πέντε αποστολές, για ε, τον καρκίνο και για τις κλιματικά ουδέτερες ευφύς πόλεις εταιρικές σχέσεις είναι κάτι που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν. Έχουμε 44 ε, τέτοιες ε, δομές στο πλαίσιο του ορίζοντα Ευρώπη, είτε θεσμικές, είτε δηλαδή δημόσιο-δημόσιο τομέα, είτε δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Έχουμε προβλέψει δύο ώρες για την ακρόαση. Κάθε ένας από τους έξι ομιλητές θα ε, έχει στη διάθεσή του το πολύ 8 λεπτά για την παρέμβασή του και έπειτα τα μέλη που θα πάρουν το λόγο θα ξεκινήσουν με τις ερωτήσεις τους αρχικά για αρχικά με τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έχουν προτεραιότητα και έπειτα θα πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι. Σας παρακαλώ να προσέξετε πολύ το χρόνο διότι πρέπει να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ε, συναδέλφους. στο τέλος κάθε ε, ενός κομματιού της ακρόασης οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο, με τους δύο προσκεκλημένους που θα μας μιλήσουν για τις αποστολές και να ξεκινήσουμε αμέσως μετά με τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων και ερωτήσεων από τα μέλη της Επιτροπής. Θα ακολουθήσει λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων και μετά θα ακολουθήσει δεύτερο, η δεύτερη σένς με τους ε, τέσσερις προσ, επόμενους προσκεκλημένους και στη συνέχεια με το δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τα μέλη της Επιτροπής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις αποστολές. Η καθηγήτρια Κριστίν Σομιέν θα λάβει πρώτο το λόγο, αντιπρόεδρος της ε, Διοικητικής Ομάδας για τον Καρκίνο από το Παρίσι. Η αποστολή αυτή αφορά όλους τους πολίτες και η κυρία Σομιάν είναι υπεύθυνη για το κομμάτι του ορίζοντα Ευρώπη που αφορά το περιβάλλον και την υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει μεγάλη προσέλευση στην Επιτροπή. Είμαστε πολύ ε, ευτυχείς που σας έχουμε εδώ για να μας παρουσιάσετε το έργο της ε, Επιτροπής. Θα σας δώσω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία. Το μικρόφωνο παρακαλώ να ανοίξετε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω καλημερίζοντάς σας εκ μέρους όλης της ομάδας μας και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσουμε το μέχρι τώρα έργο μας. Αν προλάβουμε, στο τέλος θα αναφερθώ και στις προκλήσεις και τις ανάγκες που έχουμε για το μέλλον. Γιατί λοιπόν ε, ασχολούμαστε με τον καρκίνο, διότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Εδώ σας ε, δείχνω δύο εικόνες, οι νέες ε, διαγνώσεις περιπτώσεων καρκίνου αναμένεται να αυξηθεί πάνω από το 20% στην Ευρώπη μέχρι το 2035. Και ο καρκίνος προβλέπεται να είναι το πρώτο αίτιο θανάτου στο 2030. Για να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να αλλάξουμε ε, πορεία και ο ορίζοντας Ευρώπη είναι το κατάλληλο μέσον ε, μέσω της, ε, του προγράμματος για τον καρκίνο και το αντίστοιχου σχεδίου δράσης. Αυτή η αποστολή θα συνοδεύεται από δύο επιπλέον μέτρα στο πλαίσιο του ορίζοντας Ευρώπη. Οι πέντε τομείς της ε, αποστολής μας αυτής είναι αρκετά διαφορετικοί. Ο τομέας που αφορά τον καρκίνο θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με τους υπόλοιπους ε, τομείς ενδιαφέροντος. Για, στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν μέλη, ε, υπάρχουν δύο ε, πρόεδροι, εγώ και αντιπρόεδρος και 15 μέλη ε, που αποτελούνται από εμπειρογνώμονες όλων των τομέων, από επιστήμονες, ε, βιολόγους, ακτινολόγους, εκπροσώπους ε, βιομηχανίας, παιδιάτρους που ασχολούνται ε, με τον παιδικό καρκίνο, ενώσεις ε, ιατρών, μη κυβερνητικέ οργανώσει και διεθνεί οργανισμούς. Επίσης, ε, έχουμε συνελεύσεις. Στι συνελεύσεις δεν συμμετέχουν πάνω από 30 μέλη. Η δική μα συνέλευση αποτελείται από 26 μέλη που έχουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος ο καθένας. Η συνέλευση αυτή παρέχει ένα βήμα όπου ακούγονται πρόσθετες ιδέες, όπου συγκεντρώνονται ε, εμπειρογνώμονες και όλα αυτά προς όφελος των πολιτών. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι κάτι που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Το χρονοδιάγραμμά μας εξαρτάται από την ε, προσέγγιση που υιοθετεί η αποστολή. Θα ήθελα λοιπόν να σας το παρουσιάσω. Γιατί δημιουργήθηκαν αυτές οι αποστολές. Καταρχάς για να κατευθύνουν την ε, έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη έτσι ώστε εκείνη να λύσει τις ε, προκλήσεις που ε, απασχολούν την κοινωνία και να δώσουν αποτελέσματα για τους πολίτες. Επίσης για να, συμμετέ... για να παροτρύνει τους πολίτες και τους διάφορους φορείς να συμμετέχουν περισσότερο στις διάφορες ερευνητικέ προτεραιότητες. Προτεραιότητες που θα οδηγήσουν σε καλύτερη και βελτιωμένη πρόσβαση για όλους σε αυτήν την ε, πρόσβαση, της, ε, την εμπειρογνωμοσύνη και τους ε, πόρους. Η αποστολή λοιπόν θέτει συγκεκριμένους στόχους μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χρειάζεται να ακολουθούμε συγκεκριμένη μέθοδο έτσι ώστε να αξιολογούμε τον αντίκτυπο των επενδύσεων. Και αυτό θα βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την αξία των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία και στη συνέχεια να οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα μετά από πέντε μήνε ε, συνεργασία ε, στο Συμβούλιο για τον Καρκίνο έχουμε καταλήξει μια συνένεση για τους στόχους μας. Ο στόχος ο κύριος είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να διασφαλίσουμε ποιοτικέ συνθήκε συνθήκες ζωής για τους πολίτες. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει συγκεκριμένε δράσεις σε τέσσερι τομείς. Ε, αυξημένη γνώση, πρόληψη, βελτιστοποιημένε θεραπείες και καλύτερη ποιότητα ζωή τα μέλη της Επιτροπής ε, Ήτρε γνωρίζω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την έρευνα και την ε, καινοτομία. Ε, όχι μόνο η καινοτομία οδηγεί στην απόκτηση γνώσης, αλλά βελτιώνει την ποιότητα ζωής και εδώ αναφέρομαι στην έρευνα όλων των ειδών. Επίσης, έχουμε εντοπίσει ορισμένες γκάρσιες δράσεις οι οποίες θα ωφελήσουν όλους. Φυσικά χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο οικοσύστημα γύρω μας και στην ε, καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει τις δράσεις μας ε, να διέπει η, προ... η ίση πρόσβαση, η ίση πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις, η ίση πρόσβαση στη θεραπεία, η ίση πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτά όμως ε, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς καινοτομία, που μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Και αυτό σε διεθνές επίπεδο. Θα τελειώσω με το χρονοδιάγραμμα λέγοντας ότι από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2020 θα ολοκληρωθεί το brainstorming που κάνουμε και θα καταρτήσουμε τον κατάλογο ε, που θα αποτελέσει βάση για συζήτηση με τις προκλήσεις και τις δράσεις. Σε πρώτο στάδιο θα γίνει η συνέλευση της ε, ομάδας μας στο τέλος αυτής της εβδομάδας και στη συνέχεια το Φεβρουάριο. Επίσης, ξεκινήσαμε ήδη να συναντιόμαστε με επιτρόπους, ε, με την ε, κυρία Γκάμπριελ για παράδειγμα και αυτό ήταν πολύ ε, σημαντικό για μας. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε τακτική επικοινωνία. Υπάρχουν και οι διάφορες υποομάδες, η υποομάδα για τον καρκίνο στο Συμβούλιο και άλλες, οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία και με όλους τους μπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε οι δράσεις να ε, καθοριστούν ε, σαφώς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Εδώ να πω ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία και με τις διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος, την ε, ομάδα των Ευρωβουλευτών κατά του καρκίνου, για παράδειγμα, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των ε, ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να ε, ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του τελικού εγγράφου μας που θα γίνει τον Απρίλιο στις Ευρυξέλλες. Ήδη έχουμε αρχίσει ε, κάποιες προκατακτικές συναντήσεις. Θα ξεκινήσουμε ε, πιο δυναμικά το Μάρτιο και θέλουμε να πάμε σε όλα κρατημέλη έτσι ώστε να ακούσουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες σε κάθε κράτος μέλος. Ποιε είναι οι προτεραιότητες των πολιτών στη μάχη κατά του καρκίνου. Στο Συμβούλιο έχουμε προβλέψει κάθε μέλος του να λειτουργεί ως πρεσβευτής τουλάχιστον μίας ή δύο χωρών. Τέλος, οι προκλήσεις και οι δεσμεύσεις μας. Όλοι οι εμπειρογνώμονες και στην συνέλευση και στο Συμβούλιο θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ελπίζουμε μέσα σε λίγους μήνες να καταφέρουμε να βρούμε δράσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα. Η έρευνα και η ανάπτυξη χρειάζονται 10 έως 20 χρόνια για να μπορούν να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τα κράτη-μέλη επίσης έχουν κάνει πάρα πολλά για να καταπολεμήσουν ε, αυτή την ασθένεια. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχουν εθνικά προγράμματα. Αλλά για να γίνει πραγματική αλλαγή θα χρειαστεί συγκεκριμένη δέσμευση έτσι ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καθηγητρία Σομιάν. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις και παρατηρήσεις ε, στα όσα είπατε. Αμέσως μετά τη δεύτερη παρουσίαση δίνουμε το λόγο στο δεύτερο ομιλητή από άλλον τομέα ε, αποστολής, ε, τον κύριο Emmanuel Forest, για τις κλιματικά ουδέτερες και ευφυείς πόλεις. Να μας δώσει μια διαφορετική οπτική γωνία για ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εξώτημα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάζω ενώπιόν σας ε, την ε, αποστολή μας. Ε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την αποστολή το Σεπτέμβριο, είπαμε ότι εδώ το διακύβευμα δεν είναι μόνο η έρευνα, αλλά η ανάγκη να, έχουμε, να παραδώσουμε δημόσια αγαθά στους πολίτες. Εμείς θέλουμε να παραδώσουμε 100 κλιματικά ουδέτερες ε, πόλεις μέχρι το 2030 από και προς τους πολίτες. Στο σχέδιο έκθεσης που ε, δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο, αυτά που αναφέραμε και αυτό ήταν ο τίτλος μάλιστα εμείς θέλουμε να αποδείξουμε ακριβώς ε, την ε, ορθότητα της έννοιας ε, της Πράσινης Συμφωνίας, γιατί θέλουμε να έχουμε μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα τέτοιο πιλωτικό έργο μέχρι το 2030. Αυτό βέβαια είναι κοινή πρόκληση για όλε τι ευρωπαϊκέ πόλει να βρουν λύσει στο θέμα τη κλιματική ουδετερότητα, προσαρμοσμένα πάντα στι ε, τοπικέ ιδιαιτερότητε, από το βορρά μέχρι τον νότο, από την δύση μέχρι την ανατολή ε, και με βάση και την ε, πολιτιστική κληρονομιά μα. Μια πόλη μπορεί να είναι πόλη βέβαια, μπορεί να είναι μια γειτονιά, περιοχή, ζώνη ειδικού ενδιαφέροντος όπως ένα αεροδρόμιο, μια πανεπιστημιούπολη, ένα νοσοκομείο, μια γειτονιά μιας πόλης. Το πιο σημαντικό είναι τελικά να έχουμε 100 οντότητες που θα είναι κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας ε, εν ώψη του 2050. Προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε μέσω κλιματικών συμβάσεων με τις πόλεις. Θα θέλαμε δηλαδή ε, να συνεργαζόμαστε με, με κάθε πόλη συγκεκριμένα του κάθε κράτους μέλους ε, σε ένα πνεύμα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, όλους, ε, τους, όλα τα μπλεκόμενα μέρη στο τοπικό επίπεδο για να εντοπίσουμε κενά πολιτικής και εφαρμογή της και να προσδιορίσουμε τη διακυβέρνηση, το νομικό και οικονομικό πλαίσιο και να οριστικοποιείται το έργο. Αυτή η σύμβαση θα είναι ένα μνημόνιο κατανόηση ε, μεταξύ πόλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτου μέλου και εμπλεκομένων φορέων. Και μετά θα έχουμε και εκτελεστικές ε, συμβάσεις, όπως ε, βλέπετε σε μεγάλα έργα παραχώρησης και κατασκευών. Από ποιον και για ποιον, λοιπόν. Κλιματικά ουδέτερε πόλει, είπα ότι είναι ο τίτλο, από και προ του πολίτε. Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν, η εμπλοκή ε, και συνεισφορά των πολιτών. Θα πρέπει εδώ να βλέπουμε τον πολίτη όχι μόνο σαν ε, ψηφοφόρο, αλλά σαν ε, ενεργό μέρος που θα είναι και καταναλωτής, χρήστης, παραγωγός, κάτοχος θα έχουμε πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω και όραμά μας είναι ο κάθε πολίτης να μπορεί να λέει κατανοώ ότι το κλίμα είναι σε μικρό βαθμό ε, στον έλεγχό μου και αν σε χίλια χρόνια οι άνθρωποι είναι ευτυχείς θα έχω ένα μικρό μερίδιο της ευθύνης. Αυτό είναι από το Θεό Βάνια, ένα θεατρικό έργο του ε, Τσέχοφ που γράφτηκε πάνω από 100 χρόνια πριν. Μετά περνάμε στα οικονομικά και τεχνικά μέσα. Το οικονομικό σκέλος θα αναφέρω γιατί συνήθως είναι το πιο σημαντικό. Και εσείς κύριε Πρόεδρε είπατε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε έναν ε, ε σωστό προπολογισμό. Ορίζον Ευρώπη βέβαια για την έρευνα και την καινοτομία για να έχουμε τις καλύτερες τεχνολογίες, τις κατάλληλες διαδικασίες, για να έχουμε και τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Αλλά και οι πόλεις θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα έργα και να γίνουν κλιματικά ουδέτερες. Αυτό απαιτεί επενδύσεις. Δεν θα διατρέξω όλα τα διαθέσιμα ε, δημοσιονομικά μέσα. Σίγουρα υπάρχουν τα διαθετικά ταμεία, επενδυτικά ταμεία, το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης είναι απαραίτητο φυσικά να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ε, Δύσης και Ανατολής, να υπάρχουν πιλωτικά έργα σε όλα τα κρατημέλη, ενδεχομένω. και η Πράσινη Τράπεζα, θετική εξέλιξη κατά την κατάρτιση της έκθεσής μας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και την υφιστάμενη γνώση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά για να συγκεντρώσει γνώσεις για την καινοτομία και για τα κτίρια, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είδαμε τέτοιες προσπάθειες. Ευρωπαϊκές πράσινες πρωτεύουσες, συγκεκριμένα σχέδια καθαρής ενέργειας, 100 τέτοιες ε, πιθανές ε, τοποθεσίες ε, κλιματικής ουδετερότητας. Και βέβαια Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση ε, καινοτομία για τις ευφυείς πόλεις και κοινότητες. Και μια, ε, για ένα κοινό εγχείρημα ε, για το υδρογόνο που σίγουρα θα μας απασχολήσει. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις φυσικά θα διαματήσουν σημαντικό ρόλο και για την αναδρομική εφαρμογή ε, όλων ε, των απαραίτητων μέτρων. Εκεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τον Φεβρουάριο έχουμε συνάντηση με ε, εκπροσώπους των κρατών μελών, εμπειρογνώμονες και τη συνέλευσή μας. Θα έχουμε μία υποομάδα ή επιμέρους υποομάδες που θα προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενο των συμβάσεων πώς θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμόζονται, γιατί πρόκειται για μια καινούρια έννοια. Χρειαζόμαστε βέβαια κριτήρια, διαδικασίες, ε, προϋποθέσεις, επιλογής των 100 ε, αυτών ε, μελλοντικών πράσινων πόλεων. να έχουμε πάντα κατά νου τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και από κοινού και με τα άλλα συμβούλια των υπολείπων αποστολών τέσσερις ε, ε, προσδιορίζονται ε, στο, στην Πράσινη Συμφωνία, αλλά σαφώς και εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε και, την, και τον αγώνα κατά του καρκίνου. Φυσικά και θέλουμε να εργαστούμε αποκινούμε τους συναδέλφους μας από τις υπόλοιπε συμφωνίες, και αποστολές μάλλον. Και θέλουμε και σε διεθνές επίπεδο να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία για να πετύχουμε το στόχο μας μέχρι το 2050 για κλιματική ουδετερότητα, μπορεί να είμαστε και οι μόνοι που θα πετύχουμε αυτό το στόχο πλήρως. Κλείνοντας, διάβασε ένα σχέδιο ψηφίσματος μια πρόταση να έχουμε έναν πρέσβη για το κλίμα. Αυτό ήθελα να πω, να μιλήσω για την ε, ε, κλιματική διπλωματία. Ελπίζω ε, να είμαστε κι εμείς καλοί πρεσβευτές ε, ως Συμβούλιο και είμαστε η θέση σας για ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σχόλια και παρατηρήσεις τώρα από τα μέλη. Οι δύο εισηγητές θα μιλήσουν πρώτοι. Και θα έχουμε και άλλους συναδέλφους, σκιώδεις και όχι μόνο, που θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Νίκα. Υπεύθυνος εισηγητής για τον κανονισμό. Aș vrea să θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σομιέν και τον κύριο Φορέστ για τις παρουσιάσεις τους. Και θα ήθελα δημόσια να σας ευχαριστήσω για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συνεργασία Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του προγράμματος ε, Horizon Ευρώπη, Ορίζοντας Ευρώπη. Σας ευχαριστώ που μας δείξατε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλύτερα για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Θα θέλαμε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο να στεφθεί από επιτυχία και να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες, τη βιομηχανία και να και γι' αυτόν τον τρόπο η συμβολή των ε, αποστολών, ε, των missions και των ε, εταιρικών σχέσεων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι αποστολές αναφέρονται στο κεφάλαιο παγκόσμιας προκλήσεις, αλλά θα μπορούσαν να αφορούν και άλλες συμπληρωματικέ δράσεις και άλλα συμπληρωματικά προγράμματα. Στις συνεδριάσεις με τους κοιόδης εισηγητές για τον ορίζοντα Ευρώπη πάντα θέτουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Πώς επιλέγησαν οι αποστολές, πώς λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι αποστολές θα έχουν σαφή κατεύθυνση, ε, σαφείς στόχους, ε, σαφές χρονοδιάγραμμα και σαφή προϋπολογισμό. Ε, ποια η σχέση ανάμεσα στις εταιρικές σχέσεις και στα κλάστερ. Τα κλάστερ θα βοηθήσουν τις αποστολ, ας πούμε, την αποστολή για τον καρκίνο. Και επίσης, ε, το κλάστερ για την υγεία πόσο διοργανώνει τις προκήρυξεις υποβολής ενδιαφέροντος. Πώς ε, καθορίζουμε την εταιρική σχέση στα πλαίσια μιας αποστολής. Πώς διαλέγουμε τις αποστολές στα, στα πλαίσια του προϋπολογισμού, μια και δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει για τον προϋπολογισμό. Ακόμα και αν θέλουμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Δεδομένως της συζήτηση για τη νέα στρατηγική για την Πράσινη Συμφωνία και τα νέα στοιχεία του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα που θα συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είχα, ε, η τελευταία συνάντηση με τον Ζαν Ερικ Πακέ είχε πει ότι το Climate Europe έχει τα πιο προχωρημένα έργα. Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Νίκα. Πολλές ερωτήσεις. Κάποιες uh, από αυτές όμως αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι που τις θέσατε τις περισσότερες ερωτήσεις, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες και δεν έχουμε και πολλές λεπτομέρειες, οπότε ε, ό,τι διευκρίνηση μας δοθεί θα μας βοηθήσει. Ο κύριος Έλλερ δεν είναι απλώς συντονιστής του ΕΛΚ, αλλά είναι και υπεύθυνο εισηγητής για το πρόγραμμα αυτό, Ορίζοντα Ευρώπη. Έχετε δύο λεφτά κύριε Έλλερ. Θα ήθελα να σας πω ότι το στομάχι μου δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και θέλω να δηλώσω λοιπόν ότι όσο δεν έχουμε για το στρατηγικό πρόγραμμα συμφωνία με το Συμβούλιο, ούτε προϋπολογισμό, ε, είχα ανάγκη να το δηλώσω αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Ε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση για το, στον Περκίνο. Εμείς είχαμε πει ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και τον καρκίνο και να δώσουμε έμφαση στον καρκίνο, αλλά και σε, σε ξεχασμένες ή ας πούμε άλλες αρρώστιες που δεν τις ε, έχουμε λάβει υπόψη μας με στιγμής και τις έχουμε παραμελήσει. Επίσης, ε, μπορεί τα νούμερα να είναι το 10% του προπολογισμού του δεύτερου πυλώνα. Ε, για όλες τις αποστολές θα έχουμε 750 εκατομμύρια το χρόνο. Όμως, Ίσως επειδή είμαι Γερμανός τα λέω τώρα όλα αυτά. Αλλά ποια είναι η αναλογία ε, και η χρηματοδότηση των αποστολών. Αυτή η χρηματοδότηση για τις αποστολές ε, είναι σχετικά χυμή, ενώ στον ορίζοντα 2020 ε, ξοδέψαμε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τις προκλήσεις υγείας και για έργα για τον καρκίνο. Ε, ποια είναι, εδώ έχουμε και προϋποθέσεις, ε, ε, ενώ έχουμε... Τι, τι, τι αναλογία, η αναλογία αυτών των project, ποια είναι σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ μικρός. Επίσης, μας είπατε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι νέα είναι καινούργια λεφτά μάλλον. Έχουμε 4 δισεκατομμύρια για τις έξυπνες πόλεις σε ένα κλάστερ όπου ε, τα περισσότερα λεφτά ε, πάνε για τις έξυπνες πόλεις για τη μείωση του διοξιδίου του, του άνθρακα. Ε, εδώ όμως υπάρχει χρηματοδότηση από πολλούς πόρους. Επίσης, τι θα γίνει με το κονδύλι του δεύτερου πυλώνα. Μονίμως αλλάζει. Με, μου δημιουργεί μια νευρικότητα αυτό. Επίσης, κάτι για τα διαφορετικά ταμεία, ε, με το οποίο δεν συμφώνησε το Συμβούλιο. Ε, το Ταμείο Μετάβασης δεν ε, χρησιμοποιείται για τη μείωση του του άνθρακα στις έξυπνες πόλεις. Κάθε φορά αναφερόσαστε στις διάφορες πηγές που έχουμε, αλλά οι πηγές είναι δεδομένες, δεν μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε. Δεν αυξάνονται και πληθύνονται τα λεφτά. Ε, αυτή η ομαδική χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση από διάφορες πηγές δηλαδή, ε, πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ε, στο παρελθόν έχουμε ξοδέψει λεφτά για τον καρκίνο. Αυτά τα 4 δισεκατομμύρια τα είχαμε για τις έξυπνες πόλεις. Ε, την τελευταία, περίοδο. Το πρόβλημα είναι ότι λέμε διάφορα πράγματα, πολύ φιλόδοξα, αλλά δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Τζαβάλοβα, ε, συντονίστρια του Ουρινιού. Ευχαριστώ για την ε, ακρόαση αυτή. Έχουμε εδώ πέρα ε, συντονιστές, ε, εισηγητές ε, και σκιώδες εισηγητές. Έχω, θέλω να μιλήσω για μια γενικότερη ανησυχία για την επιτυχία των αποστολών. Θέλω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβω το με, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον και αν θα υπάρχει περίπτωση επιτυχίας. Ε, υπάρχουν μη επιτυχημένες αποστολές, ας πούμε, που δεν έχουν υλοποιήσει τους στόχους τους. παρόλα αυτά είναι υποφελής για τους πολίτες λόγω των ε, δευτερογενών επιπτώσεων οικονομικών, ε, στην υγεία κτλ. Ε, όμως ε, συχνά οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι πόροι έχουν επενδυθεί για κάτι τέτοιο. Ας πούμε, για να είναι πετυχημένος ορίζοντας Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενήμερη όλη η κοινωνία για τις αποστολές θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ περισσότερο η επικοινωνία. Δεν μπορούμε να χάσουμε καμία ευκαιρία για να φτάσουμε στους πολίτες, για να τους ε, κοινωνήσουμε αυτό τον ενθουσιασμό στο project αυτό ε, και να τους δείξουμε τις αλλαγές που κάνουν ε, αυτά τα project ε, καινοτομίας και έρευνας. Θα πρέπει όλοι οι φορείς να εμπλακούν, να είναι έτοιμοι να απορροφήσουν, να, να δεχτούν ας πούμε αυτές τις ε, θετικές επιπτώσεις. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένα παραδείγματα από τους εκπροσώπους των δύο αποστολών που πήραν το λόγο. Από τους πράσινους έχουμε την κυρία Τζίνα Ντάουντιν. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συναντηθήκατε μαζί μα. Ε, χαιρόμαστε για τι πληροφορίε που μα δώσατε, και την ανταλλαγή πληροφοριών και να δυνατότητα να ακούσουμε κάποιε απαντήσει ερωτήσει μα. Οι αποστολέ και οι εταιρικέ σχέσει θέλουμε όχι μόνο ε, να έχουν αποτελέσματα για να λυθούν οι προκλήσει, αλλά θα λάβουν και δισεκατομμύρια για να εφαρμοστούν. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και η σωστή εφαρμογή και επίπεδο διαφάνεια επαρκέ. Μία ερώτηση προ τον κύριο Φόρεστ για, την, ε, για τις έξυπνες ε, πόλεις και κλιματικά ουδέτερες. Ε, τις επόμενες δεκαετίες στη φιλία θα, θα ε, επιδεινωθεί. Άρα ε, είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό το κομμάτι για τις έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Από την άλλη ξέρουμε, ε, λιγότερες, λιγότερα αυτοκίνητα σημαίνει λιγότερες εκπομπές, λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, καλύτερος αέρας και καλύτερο περιβάλλον. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι έργα υπό αυτό το κομμάτι αποστολής θα αντιμετωπίσουν ε, τα κενά που έχουμε στην γνώση για να πετύχουμε πραγματικές λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των αστικών περιοχών. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι συγκεκριμένα project σε αυτό το κομμάτι αποστολής συνεισφέρουν στην μείωση των εκπομπών και πώς θα το μετρήσουμε αυτό το πράγμα, αυτή την επίπτωση. Τι μέτρα θα εφαρμόσετε για να εξασφαλίσετε ότι οι αποστολές αυτές οδηγούν σε λύσεις ε, χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, για τη συμμετοχή των πολιτών, μετά από αυτά που είναι οι συνάδελφοι, τι κάνατε ή τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε αυτή την άμεση αλληλεπίδραση με τους πολίτες ε, και ομάδες εκπροσώπων για να επιλέγετε, όταν επιλέγετε τα project ε, στον τομέα της αποστολής σας. Π.χ. ανθρώπους ε, που έχουν ε, διαφορετική κινητικότητα ή περιορισμένη κινητικότητα. Μια σύντομη ερώτηση προς την κυρία Κομιέν για τον καρκίνο, την αποστολή για τον καρκίνο. Τα projects αυτή την αποστολή πώς θα εστιάσουν προς ένα κοινό στόχο να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, να προλάβουν το να ξοδεύουμε πόρους με λιγότερο στρατηγικό τρόπο για τις διάφορες προτεραιότητες. Η κυρία Λίτζη, ε, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη 100 δισεκατομμύρια ευρώ και το Συμβούλιο θα μειώσει αυτό το ποσό. Και έχουμε μία συζήτηση ήδη και μία διελκυστήνα στα πλαίσια του Πουδουπού. Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι κατά πάση, πάσα περιπτώσει από τα πέντε μίσον στο στρατηγικό σχέδιο δεν θα δρομολογηθούν και οι πέντε αποστολές αυτές ταυτόχρονα. Το γεγονός ότι σήμερα είναι παρόντες ε, οι εκπρόσωποι του, της αποστολής ε, καρκίνος και έξυπνες πόλεις μπορεί να σημαίνει ότι οι επόμενες τρεις αποστολές θα ξεκινήσουν μετά το 2024 ή τυχαίο είναι αυτό που είσαστε οι δύο μόνο εδώ. Και έπειτα, μπορείτε να εκτιμήσετε τις οικονομικές ανάγκες απαραίτητες και τα απαραίτητα χρήματα για να υλοποιήσετε τα προκαθορισμένα αποτελέσματα είναι οριζόντιο ερώτημα αυτό. Ε, στο σχέδιο, το νομικό σχέδιο για τον ορίζοντα Ευρώπη, ε, οι αποστολές θα πρέπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φτάσουν σε ένα προσμετρήσιμο στόχο, έτσι λέγεται, και να έχουν επίπτωση στην κοινωνία μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας και οι επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να είναι σημαντικές για ένα σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού ε, πληθυσμού και γενικότερα, πιο συγκεκριμένα με βάση την, ε, το αντικείμενο της αποστολής, αλλά και γενικότερα για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Το Συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει την κλίμακα των ε, στόχων των αποστολών. Αλλά επειδή έχουμε και συγκεκριμένα, ας πούμε, συγκεκριμένους στόχους, έχετε τα mission board. Ε, τα συμβούλια αυτά θα είναι πραγματικά ανεξάρτητα ή απλώς θα υλοποιούν τη θέληση της Κομισιόν ή ακόμα χειρότερο, ε, μόνο την πολιτική βούληση εκείνων που βρίσκονται στα board. Με ποιον τρόπο θα λεπιδράσετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι συνομοθέτης και που θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, ζητώ όπως κι άλλοι απόλυτη διαφάνεια, ούτω ώστε να ξέρουμε τι αλληλεπίδραση θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα συμβούλια των αποστολών. Γιατί στην πραγματικότητα ο συνομοθέτη θα πρέπει να επιλέξει, να συνεπιλέξει το δρόμο για τη συγχρηματοδότηση. Ή για τη, συγγνώμη, για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τασονόφσκι για το CCR. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε λεπτομέρειες για αυτούς τους δύο τομείς. Με τους συναδέλφους μου συζητούσαμε όλο το νομοθετικό πακέτο του ορίζοντα. Δεν ήταν εύκολο. Γνωρίζαμε πως θα είχαμε αρκετή πίεση για τα οικονομικά. Οι συνάδελφοί μου το ανέφεραν εξάλλου. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδεθούν αυτά τα προγράμματα με άλλα, για παράδειγμα τις εξύπνες πόλεις. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν περιμένετε ε, χρηματοδότηση και για άλλα προγράμματα όπως το Γαλιλαίος ή το Κοπέρνικος. Νομίζω πως ε, θα μπορούσαν να από πολύ χρήσιμα. Επίσης και λόγω των δεδομένων που θα έχουν στη διάθεσή τους και ιδιαίτερα μάλιστα αν συνδεθούν με τις έξυπνες πόλεις. Διότι ανησυχώ πως αν ε, τα εξετάσουμε μεμονωμένα, τα προγράμματα αυτά δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν συνέργειες. Και δεν θα επιτύχουν σε τελική ανάλυση το στόχο τους. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια πόλη που θα έχει βρει μια λύση και δεν θα μπορεί να βοηθήσει ε, αν δεν είναι συνδεδεμένη. Γι' αυτό θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να είναι πανευρωπαϊκό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμπεριλαμβάνεται και το θέμα του καρκίνου, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει αρκετά Ε, για τον παιδικό καρκίνο βέβαια δεν ξέρω ε, τι θα γίνει. Θα δώσω το περισσότερη έμφαση εκεί. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις ε, συνδέσεις με τα άλλα project. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στις πέντε παρεμβάσεις των άλλων συναδέλφων. Εδώ προτείνω να μιλήσετε μόνο για ένα λεπτό ο καθένας, έτσι ώστε οι εμπειρογνώμονες να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν για πέντε λεπτά και για να προλάβουμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Δεν θα κάνω την ερώτησή μου για τις ε, εταιρικέ σχέσεις, διότι δεν ε, ήμουν εδώ. Δυστυχώς θα μιλήσω μετά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τόια. Ένα λεπτό. Καταρχάς σας ενθαρρύνω και σας στηρίζω τις αποστολές. Θα είμαστε στο πλευρό σας στο Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον ε, εξ ονοματός μου μιλάω. Δεύτερο, περιεχόμενο και μέθοδος. Στο παρελθόν δεν υπήρχε συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο, σε διασυνοριακό επίπεδο για την έρευνα. Και αυτό μείωσε τις προσπάθειές μας και την επίπτωσή τους. Χωρίς συνεργασία κάθε κράτος δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε τους πόρους για να έχουμε και μετρήσιμους υλοποίηση των στόχων, μετρήσιμοι. Γιατί καλό είναι να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που έχουμε προσπαθήσει τα κράτη-μέλη να κάνουν μόνα τους σε επίπεδο κλάστερ. Είναι θέμα συγκέντρωσης. Μόνο έτσι φτάνουμε σε κρίσιμη μάζα. Έχω λίγα δευτερόλεπτα για το περιεχόμενο. Αυτή η αποστολή για τον ε, καρκίνο ε, ξεκίνησε από την καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου. Το θυμάμαι εγώ πάρα πολύ καλά. Και μετά επεκτάθηκε. Θα ήθελα ο παιδικός καρκίνος, που είναι ο πρώτος, ε, η πρώτη σκοτόστρα στην Ευρώπη, στην ε, Ήπειρό μας, να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχάσουμε ότι έχει προτεραιότητα ο παιδικός καρκίνος ε, στα πλαίσια της αποστολής αυτής, του μίσον αυτού. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ισάψ από το Ρινιού. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση και για τους ε, δύο προσκεκλημένους και για τις δύο αποστολές δηλαδή. Καταρχάς, ό,τι αφορά την συμπερίληψη των πολιτών, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται ο ρόλος τους σε αυτές τις αποστολές. Ε, μου φαίνεται πως ε, θα υπάρχουν διαφορές στις δύο αυτές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, ο οποίος είναι και περιορισμένος από όσο ακούω. Ε, η πρωτοβουλία των ε, έξυπνων κλιματικά ουδέτερων πόλεων ίσως χρειάζεται ε, να ιεραρχηθεί διαφορετικά από την πρωτοβουλία για τον καρκίνο. Ο καρκίνος θέλει έρευνα, θέλει στοιχεία. Αναφερθήκατε και στην ε, πρωτοβουλία ε, που υιοθέτησε η κυβέρνηση Ομπάμα, δηλαδή τον ε, χάρτη για τον καρκίνο. Οπότε θα με ενδιαφέρε να δω πώς το συνδέεται. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάλβες Μουνιός. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι στηρίζω αυτές τις αποστολές. Θεωρώ όμως πως αυτές οι αποστολές θα πρέπει να έχουν απήχηση, θα πρέπει να ξεκινήσουν και να εφαρμόζονται. Η κυρία Τόγια είπε ότι Η κυρία Τόγια είπε ότι πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα με τον παιδικό καρκίνο. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα λοιπόν, ε, διότι ως συνομοθέτες είναι βασικό να γνωρίζουμε όσο περισσότερα μπορούμε για αυτό το εγκάρσιο ζήτημα. Μετά, πώς μπορούμε να συνδέσουμε την ε, ψηφιακή μετάβαση και την ασφάλεια. Τέλος. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για αυτά τα κριτήρια επιλογής και την διαδικασία, δηλαδή πώς θα διαμορφωθούν, με βάση ποια κριτήρια θα επιλέγετε τα project και αν έχετε σκεφτεί την ε, δυνατότητα αλλαγής προτεραιοτήτων ανάλογα την τοποθεσία, ανάλογα το μέρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόλης Περέζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τον κύριο Φόρες την ερώτηση. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή ε, για, πάνω στην νομοθεσία που θα διέπει το Ευρωπαϊκό ε, Ινστιτούτο Καινοτομίας. Θα έχουμε ε, ειδικέ εταιρικέ σχέσεις εκεί. Στα πλαίσια του κλίματος, πώς θα συνεισφέρει η δουλειά αυτής της εταιρική σχέσης και της αποστολής που εκπροσωπείτε εσείς υπέρ της κλιματικής ουδετερότητας των έκθων πόλεμων πόλεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο των σφιχτών προϋπολογισμών και των χρημάτων που δεν έχουν άφθονα τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά εργαλεία για ίδια ε, project. Το θέμα είναι να υπάρχουν συνέργειες και συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ε, τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ξεκινάμε με σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και στην αρχή, ήταν πολύ σημαντικό για μας ως μέλη του Συμβουλίου των Αποστολών να ακούσουμε τις ε, προθέσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μοδοποιήσω τα σχόλια σε τρία τμήματα. Πρώτο και πολύ σημαντικό για μας είναι η εμπλοκή των ε, πολιτών. Παρότι έχουμε να κάνουμε εδώ με τον καρκίνο και έχουμε συνηθίσει να συνεργαζόμαστε με συλλόγους ε, εκπροσώπησης ασθενών και γονέων. Παρ' αυτά δεν έχουμε ακόμα συνηθίσει να συνεργαζόμαστε με πολίτες ευρύτερα. Ο καρκίνος πρέπει όμως και η καταπολέμηση του καρκίνου πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες. Εάν θέλουμε πραγματικά να ε, ωφελούνται οι πολίτες από την έγκαιρη διάγνωση και, τον, και τους διαγνωστικούς ελέγχους κατά του καρκίνου, πρέπει να κάνουμε περισσότερα μπορεί σε άλλε αποστολέ ε, η κατάσταση να είναι καλύτερη ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με του πολίτε, αλλά εμεί θέλουμε πραγματικά να το βάλουμε και το ιεραρχήσουμε σαν προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι θέλουν οι πολίτες στην Εστονία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δεν είναι μία ε, συνολική και πανευρωπαϊκή ένωση πολιτών. Θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένα τι θέλουν οι πολίτες σε κάθε χώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε σε τοπικό επίπεδο και να ακούσουμε τις θέσεις των πολιτών σε κάθε χώρα. Ακόμα και στο εσωτερικό μιας χώρας ε, αλλάζουν οι απόψεις και οι προτεραιότητες από περιφέρεια σε περιφέρεια. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, στην Νίκαια, οι προτεραιότητες των πολιτών μπορούν να είναι διαφορετικές ε, από ότι σε άλλες ε, περιοχές της Γαλλίας που είναι πιο αγροτικές, ας πούμε. Γι' αυτό πρέπει να συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Δεύτερον, κάποιοι δεν ακούσατε αυτά που θα θέλατε για να επικεντρωθούμε ε, στους μικρούς αντοσογωγικών καρκίνους ή ε, τους ε, παιδικούς καρκίνους. Φυσικά και βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών μας και του ενδιαφέροντός μας. Όταν λέμε ότι θέλουμε περισσότερη γνώση, αυτό φυσικά καλύπτει ε, και καρκίνους για τους οποίους δεν έχουμε σημειώσει καμία απολύτως πρόοδο. Το μεγάλο, για το μεγάλο ποσοστό των παιδικών καρκίνων αυτό ισχύει. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά και να συγκεντρώσουμε περισσότερε πληροφορίε. Για του παιδιατρικούς καρκίνους να πω επίση ότι ε, αυτό που ανέφερα για την ποιότητα διαβίωση ε, έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με του επιζώντε καρκίνων που είναι παιδιά που αντιμετωπίζουν ε, παρενέργειες ε, σε σχέση με τις θεραπείες τις οποίες έχουν υποστεί και είναι σημαντικό και τα παιδιά και οι γονείς τους να γνωρίζουν τι να κάνουν, τα παιδιά αυτά πώς θα μεγαλώσουν ως ενήλικες και όχι σαν καρκινοπαθείς πια. Για το Blue Ribbon και για το Moonshot, να πω ότι ε, θέλουμε προγραμματισμό που αναφέρεται στις διάφορες ε, εκθέσεις και είναι ένας διαφορετικός τρόπος για μας να προγραμματίσουμε την έρευνα, πολύ διαφορετικός από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θέλουμε να έχουμε σταχευμένες δράσεις από κοινού και με τους πολίτες και με τους ε, συλλόγους ασθενών και γονέων αυτό θα μας επιτρέψει και είμαστε αισιόδοξοι να έχουμε μια σωστή εφαρμογή και σωστή κατανόηση από τους πολίτες για ε, τους στόχους που θα επιτύχουμε μέσω των ενεργειών μας. Ευχαριστούμε κύριε Φόρεστ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για ε, τις ερωτήσεις, τα σχόλιά τους. Όλα αυτά σε, μας βοηθούν να συνεχίσουμε το έργο μας. Ε, Ξεκινώ από την ε, συνεισφορά των πολιτών και αυτό που αναφέρθηκε για τα λιγότερα οχήματα που οδηγούν σε λιγότερη συμφόρηση, λιγότερη ρήπανση και το καθεξής. Όλα αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμά μας και είπαμε ότι οι μεταφορές ε, είναι πολύ συγκεκριμένη προτεραιότητα ε, της αποστολής μας. Βέβαια, το θέμα των μεταφορών δεν μπορεί να επιληθεί χωρίς διαφορετικό σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα υπήρξε μια πρόσφατη μελέτη που λέει ότι αν θέλουμε να έχουμε πλήρη επιτυχία στην ε, ε, χρήση ηλεκτρικών ε, οχημάτων, θα πρέπει να απαγορεύσουμε, απαγορεύσουμε την κατοχή και χρήση μεμονωμένων οχημάτων και αυτό θα δεκαπλασιάσει τις υποδομές για τα ηλεκτρικά οχήματα. Δεν λέω ότι αυτή είναι πρόταση. Απλώς ήθελα να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, γι' αυτό και σας ανέφερα ε, και παρέθεσα ε, τον Τσέχοφ, ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Αυτό απαιτεί καλύτερη και μόνιμη ε, επικοινωνία. Το πρώτο εξάμεινο αυτό ακριβώ θα κάνουμε. Θα επισκεφθούμε πόλεις, θα έρθουμε σε επαφή με πολίτε. να μάθουμε περισσότερα για τις εξελίξεις ε, στις πόλεις, όχι τους αρχιτέκτονες που δουλεύουν στα γραφεία τους, ε, με τον κόσμο που κυκλοφορεί στον δρόμο. Μετά για τα kicks και όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας που είναι μια τεράστια πρόκληση για μας. Να συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες, να δούμε τι υπάρχει. Και υπάρχουν πολλά. Και θέλουμε, όπως είπα, να διαμορφώσουμε αυτούς τους ε, κόμβους σε 100 διαφορετικές ε, πόλεις με το 2030. Μετά για τα χρηματοδοτικά μέσα δεν εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, να προσδιορίσω ότι η χρηματοδότηση του Ορίζοντα Ευρώπη θα επικεντρωθεί στο τμήμα έρευνας και κοινοτομίας για τη διαμόρφωση νέων ε, ε, τεχνολογιών που θα μας διευκολύνουν στο έργο μας. Για μια κλιματικά ουδέτερη Ήπειρο χρειαζόμαστε 6.000 δις για τον μετεξοπλισμό παλαιών κτηρίων, ε, την ε, αναβάθμιση ε, των υποδομών, από τα οχήματα, τα συμβατικά να πάμε σε ηλεκτρικά και ούτω καθεξής. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει πιέσεις για τον προπολογισμό. Χρειάζεται μεγαλύτερη όμως χρηματοδότηση. Τα τέσσερα δις για τις ευφυείς πόλεις αφορούσε μόνο τις ευφυείς πόλει, αλλά τα δικά μα έργα είναι ευρύτερα από τις ευφυείς πόλει και μόνο. Γιατί όταν λέμε ευφυείς πόλεις, τι εννοούμε ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών προ όφελο των πολιτών, αλλά όταν μιλούμε για κλιματικά ουδέτερη πόλη, χρειαζόμαστε πλήρη εμπλοκή όλων των φορέων και των πολιτών. Πολύ πιο σύνθετο. Για τα χρηματοδοτικά μέσα, κλείνω μια προσωπική γνώμη από την επιχειρηματική μου σταδιοδρομία, το πρόβλημα ποτέ δεν είναι να βρούμε χρηματοδότηση. Το θέμα είναι πάντα να βρούμε καλά έργα. Όταν έχουμε καλό έργο, βρίσκουμε και τη χρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, απαιτούνται και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά ελπίζουμε να, και με τη δική σας ε, στήριξη και συνδρομή να πείσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι τα ε, έργα που προτείνουμε είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο επόμενο τμήμα, εταιρικέ σχέσεις. Έχουμε δύο κοινοπραξίες, ε, μία εταιρική σχέση δημοσίου-δημοσίου και μία ε, συμβατική εταιρική σχέση ε, φορέων του δημοσίου. Πρώτο ομιλητή είναι ο Άξελ Κράιν, εκτελεστικό διευθυντή τη κοινοπραξία Καθαρή Ουρανή, που είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση στην αεροναυπηγική. 8 λεπτά ο κάθε ομιλητής, ο κάθε πανελίστας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι υπερβουλευτέ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρουσίαση υπενθυμίζοντας τι έχουμε πετύχει τα τελευταία 10 χρόνια συνολικά. Εδώ βλέπετε το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί, τα ερευνητικά όργανα, τα πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία γενικά που δημιουργούν αυτό το μοναδικό πλαίσιο, το μοναδικό οικοσύστημα που είναι πολύ αποτελεσματικό και με καλές επιδόσεις. Είναι κάτι που μας κάνει περήφανους, αλλά δεν αρκεί. Βλέπετε εδώ στην επόμενη διαφάνεια για τους περιβαλλοντικούς στόχους, για το διοξείδιο του άνθρακα ε, τα οξύδια του αζότου και τον ε, θόρυβο είναι μεταξύ 20 και 30% και με βάση τις πρόσφατες μελέτες αντικτύπου φαίνεται ότι θα τους υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, αλλά πόρο απέχουν για να συμμορφωθούμε με τους στόχους του Παρισιού και να υλοποιήσουμε την πράσινη συμφωνία που έχει διατυπώσει η Κομισιόν. Επομένω σημαντικά ωφέλη, αλλά ανεπαρκή. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Εδώ εξετάζουμε τις, την πορεία των εκπομπών ε, αερίου του, του θερμοκηπίου. Βλέπουμε την ε, καθοδική πορεία από εδώ που βρισκόμαστε, από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή το που θέλουμε να φτάσουμε ε, το 2050. Μιλάμε για μια τεράστια μείωση. Είναι τεράστια πρόκληση για να το πετύχουμε αυτό. Ειδικά για την αεροπορία που είναι τμήμα των μεταφορών, γιατί από τη μία η ασφάλεια, οι προποθέσει για την ασφάλεια είναι τέτοιε και έχουμε και προϊόντα μεγάλου κύκλου ζωή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε προσπάθειε σε επίπεδο πολιτική. Ε, όλοι οι ιδιωτικοί φορεί, τα πανεπιστήμια, οι ερευνητικοί οργανισμοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, ο κλάδο, ε, να κάνουν μαζί προσπάθεια για να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό. Του τελευταίου μήνε τι έχει γίνει. Ε, οι ιδιωτικοί φορεί, του βλέπετε εδώ, οι οποίοι δουλεύουν πάνω στο θέμα αυτό και αναπτύσσουν ένα κοινό όραμα και δεσμεύσεις. Τα, οι δεσμεύσεις λένε ναι, εμείς οι ιδιωτικοί φορείς θα πετύχουμε την, κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 αν είμαστε ενωμένοι μαζί με την Ένωση και μαζί με όλους τους συμφεροντούχους που είναι σημαντικοί γι' αυτό. Και εδώ βλέπετε όλους τους φορείς που είναι τμήμα αυτής της προσπάθειας, πανεπιστήμια, ερευνητικές οργανώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον κλάδο. Ε, εδώ βλέπετε την ΕΑΖΑ, που είναι ο ρυθμιστικός φορέας, που πιστεύουμε ότι έχει σημαντικό ρόλο, είναι σημαντικό ε, να συμμετέχει και ο φορέας πιστοποίηση από την αρχή στην όλη προσπάθεια. Κοινό όραμα, μπορούμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα και στην αεροπορία μέχρι το 2050, αλλά απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εταίρους. Τεχνολογία τώρα. τι αναπτύσσουν διάφοροι φορείς. Κοιτάμε τις ομάδες προϊόντων. Εδώ βλέπετε τα, κάθετα κλάστερ, ε, τα αεροσκάφη μεταφόρηση επιβατών, ελικόπτερα, ε, περιφερειακά αεροσκάφη, ε, τα αεροσκάφη μικρών και μεσαίων ή μεγάλων διαδρομών. Και τα οριζόντια κουτάκια μιλάνε για τις τεχνολογίες που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα κάθετα κλάστερ. Έχουμε ε, όθηση ηλεκτρική, υδροηλεκτρική, ε, τουρμπίνες, για να έχουμε βιώσιμα καύσιμα. Η συνδυασμένη προσπάθεια θα μας οδηγήσει στην υλοποίηση του 50% του στόχου. Και μαζί με τις επιχειρησιακές βελτιώσεις και με το στόχο των βιώσιμων ε, καυσίμων μπορούμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα με το 2050. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να γίνει συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια για τα διάφορα κλάστερ, ούτω ώστε οι τεχνολογίε οι οποίε αναπτύσσονται να γίνονται με βάση τα κλάστερ τα οποία περιγράφουμε. Υπάρχουν κάποιε προκλήσει ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, που αναφέρουν ιδιωτικοί φορεί. Καταρχά είναι η σύνδεση της έρευνας που να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία ε, σήμερα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και που είναι ευθύνη της ε, Κομισιόν ε, και την έρευνα που υπάρχει στα πλαίσια του πλαισίου καθαρή ουρανή. η αλληλεπίδραση αυτών των δύο, επειδή είναι διαφορετικέ προτεραιότητε, διαφορετικέ στρατηγικέ, διαφορετικέ συνδρομέ κτλ., οι αλληλεπιδράσει είναι μικρέ, περιορισμένε. Αυτό που προτείνουμε στον ορίζοντα Ευρώπη είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο πυλώνε, ε, για να, καταχάσει ένα πυλώνα για να δημιουργηθούν ιδέες, γιατί οι στόχοι είναι τόσο μοναδικοί που πρέπει πραγματικά να υπάρξουν γρήγορα νέες ιδέες και να ενσωματωθούν εν συνεχεία ε, το συντομότερο δυνατό, ούτω ώστε να πετύχουμε την ε, επίπτωση που θέλουμε στο τελικό προϊόν. Και ο συνδυασμό των δύο, δηλαδή το συνεργατικό κομμάτι και το, η επίδειξη ας πούμε του προϊόντος, ε, ή τη έρευνα, ας πούμε, χρειάζεται να γίνει. Ε, συνέχεια, συνέργεια με άλλα προγράμματα. Εδώ βλέπετε αριστερά τον ορίζοντα 2020. Είχαμε συμμετοχή διαφόρων περιφερειών σε όλη την Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν τα διαρθωτικά ταμεία. Υποστηρίζουμε τις ε, περιφέρειες, δίνουμε τεχνική στήριξη και μέσω και η στήριξη μέσω των διαφόρων προτεραιοτήτων σε τοπικό επίπεδο για να πετύχουμε ε, συνέργειες 50 εκατομμύριων ανάμεσα στα διαφορετικά ταμεία και στο, στους καθαρούς ουρανούς. Στον ορίζοντα Ευρώπη βλέπετε τελείως διαφορετικό πλαίσιο, άλλη αρχιτεκτονική. Έχουμε μια καινοτόμα αρχιτεκτονική, όπου η ολοκλήρωση των διαφόρων προγραμμάτων σε ή το πάτρεμα των προγραμμάτων ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, με μπλε, μπλε, τα μπλε συννεφάκια. Έχετε διάφορα προγράμματα. Έχετε κάτι που είναι πολύ διαφορετικό εδώ, γιατί έχετε και τεράστια χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως ε, χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαφορετικά ταμεία. Ο στόχο της κλιματικής ουδετερότητα ε, προϋποθέτει τεράστια προσπάθεια που την έχουμε αποτιμήσει σε χρήματα για το πρώτο κομμάτι έρευνα και καινοτομία <coughs> την επόμενη δεκαετία μέχρι το 28-29 η προσπάθεια έχει αποτιμηθεί σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 12 δισεκατομμύρια θα δρομολογήσουν την ανάπτυξη προϊόντων. Θα προκαλέσουν ανάπτυξη προϊόντων. Αυτό το κόστο θα το φέρει η βιομηχανία. 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τέλο είναι τα προγράμματα αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν από τι αεροπορικέ εταιρείε. Εδώ χρειαζόμαστε 5-3. 5-3. Είναι η μισή παγκόσμια αγορά. Αν η μισή αγορά, λοιπόν, ε, παγκόσμια αγορά θα διατηρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για 12 αρχικά ε, δισεκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια και μετά 5-3. Έχουμε την εταιρική σχέση καθαρή αεροπορία, που είναι το μισό του προγράμματος, το 12 δισεκατομμύριο και το υπόλοιπο μισό προέρχεται από τι συνέρχειε με, με, τα άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και με τη συμμετοχή των ε, διαφορετικών ταμείων. 2 επί 6 μα κάνουν 12 δι. Το 6 είναι μαγικό νούμερο στην εταιρική σχέση καθαρή αεροπορία, ούτω ώστε να υπάρχει μόχλευση για τι απαραίτητε επενδύσει. Κλείνω. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει το πλαίσιο τη προκλήση, μιλάει για τι προκλήσει Υπάρχει σαφής ε, φιλοδοξία από τους ποιοτικού φορείς ότι μπορεί να γίνει, να η πράσινη συμφωνία, αλλά δεν χρειάζεται εξέλιξη, χρειάζεται επανάσταση. Οι ιδιωτικοί φορείς πιστεύουν ότι η εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού είναι το εργαλείο για να γίνει αυτή η επανάσταση και να υπάρχουν επιπτώσεις. Τα επόμενα βήματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να υπάρχει σωστή το κανονιστικό πλαίσιο, σωστή χρηματοδότηση, ούτω ώστε να υπάρξουν αυτές οι συνέργειες και να θέσουμε εμείς ως Ευρώπη την παγκόσμια σκηνή και τους παγκόσμιους στόχους. Σας, σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε με ερωτήσεις. Προς το παρόν θα περάσουμε στον κύριο Μπάρτ Μπίμπικ, εκτελεστικό διευθυντή της κοινή επιχείρησης για στήλες καυσίμου και υδρογόνου. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας εξηγήσουμε ε, τι πιστεύουμε εμεί πώ θα είναι απαραίτητο για την κοινή επιχείρηση ε, στυλώνα καυσίμου και υδραγόνου. καθώς και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας. Η στήλωση καυσίμου και υδρογόνου έχουν διάφορε τεχνολογίε στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κλιματική Πολιτική, η οποία τώρα χαρακτηρίζεται από την Πράσινη Συμφωνία. Είναι αναγκαία αυτή η Πράσινη Συμφωνία, θεωρούμε, και βασικά πιστεύουμε πω ε, ο ένα χρειάζεται τον άλλον. Η δική μα συνεισφορά θα είναι η μείωση που έχουμε προτείνει. Ε, μία μείωση τη τάξη του 50-55% είναι τεράστια ε, πρόκληση και γι' αυτό χρειαζόμαστε το υδρογόνο. Η κοινή μας επιχείρηση, όπως ξέρετε, είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όμως ε, ήταν απαραίτητη για να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, αυτό το οικοσύστημα που θα φιλοξενήσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το υδρογόνο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτές οι ιδέες που χαρακτηρίζονται από καινοτομία να ε, μεταφερθούν στην αγορά. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία. Και εμείς αυτό κάνουμε. Συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους με την κοινωνία των πολιτών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απλούς πολίτες, αλλά και με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας. Οι κοινέ επιχειρήσεις επίσης στόχο έχουν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις οι μικρομισές επιχειρήσεις θα θελήσουν να επενδύσουν σε ένα μακρόπνοο σχέδιο. Ακριβώς ε, για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι εταιρικές σχέσεις, διότι η πλειοψηφία των ε, μελών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 30% της χρηματοδότησης πηγαίνει σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι κοινέ επιχειρήσεις λοιπόν δίνουν γρήγορα αποτελέσματα στους πολίτε, διότι μπορούν να δοκιμάσουν, να τεστάρουν ένα προϊόν πριν το ε, εγκρίνουν για διάθεση στην αγορά. Επίση, δημιουργούμε θέσει απασχόληση στις ε, μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις. Δίνουμε ερεθίσματα και κίνητρα για ε, περισσότερα και φροντίζουμε ε, μέσω της χρηματοδότησης που έχουμε όλοι οι μισθοί να καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της Κομισιόν. Να σας πω δύο λόγια για κάποια νούμερα. Έχουμε 263 project που χρηματοδοτούνται από 457 εκατομμύρια ευρώ. Ε, νομίζω πως ε, μπορούμε να πούμε πως είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Το υδρογόνο, τι μπορεί να προσφέρει. Το 2050 το υδρογόνο θα αποτελεί μεγάλο κομμάτι της αγοράς ενέργειας, πάνω από 20%, 24% περίπου. Μπορούμε να ε, μειώσουμε ε, να, τις εκπομπές κατά 560 μεγατόνους ετήσιο εισόδημα έως 820 δισεκατομμύρια ευρώ και να αυξήσουμε τις απασχόληση κατά 15%. Οι θέσεις όμως αυτές δεν θα δημιουργηθούν από το πουθενά. Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία. Γι' αυτό και χαρακτηριζόμαστε από τρεις πυλώνες. Πρώτον, παραγωγή υδρογόνου. Δεύτερον, ηλεκτρόλυση. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε κλίμακα μεγαβάτ. Έχουμε περάσει από τα κιλοβάτ στα μεγαβάτ και θα πρέπει να περάσουμε και στα γίγαβατ. Δεύτερος ε, πυλώνας, ε, διανομή. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες αποθήκευσης μεγάλου, μεγάλης ποσότητας ενέργειας, να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε σε αποθήκες υδρογόνου τις υπάρχουσες έπειτα, να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για να χρησιμοποιήσουμε άλλα αέρια όπως το μεθάνιο, ας πούμε. Έπειτα, ε, ο τελικός χρήστης ποιος είναι. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας. Ε, τα οχήματα ε, που θα χρησιμοποιηθεί, μεταφορές. θα συνεργαζόμαστε λοιπόν με όλους τους φορείς. Τέλος, θα χρειαστεί φυσικά να διατηρήσουμε τα πρότυπα ασφαλείας, αλλά και να ασχοληθούμε με την αλυσίδα εφοδιασμού. Ε, το, την δευτερογενή παραγωγή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης. Τι έχουμε προτείνει λοιπόν από χρηματοδότηση. 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, εταιρική σχέση καθαρό υδρογόνο. Μέχρι το 2030 Θέλουμε οι συνολικέ επενδύσει να φτάσουν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Με, από το 2021 στο 2027 τα 8,7 δισεκατομμύρια και 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ανά εταιρική ε, σχέση. Αυτή είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινή αυτή επιχείρηση επίσης θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 29 περιφέρειες όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ασχολούμαστε επίσης με την ευφυή εξειδίκευση. Βέβαια, είναι ευπρόσδεκτη κάθε περαιτέρω συνεισφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, κανονικά θα έπρεπε να τον διπλασιάσουμε, διότι μιλάμε για ε, μεγάλο project και σε όγκο και σε έκταση γεωγραφική. Ε, επίσης, ένα όχημα που κινείται με υδρογόνο για να βγει στους δρόμους θέλει περίπου 40.000 ευρώ. Είναι λοιπόν μεγάλα τα ποσά, γι' αυτό και χρειαζόμαστε διπλασιασμό του προϋπολογισμού. Τώρα, η Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ βλέπουμε ότι η Κίνα επενδύει 4 ευρώ ανά πολίτη, η Ιαπωνία 3. Στην Ευρώπη 0,5 ευρώ, 50 λεπτά ανά πολίτη. Αυτό συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη σήμερα. Έχουμε το πλεονέκτημα, το έχουμε ξεκινήσει εγκαίρως, είμαστε μπροστά σε αυτή την τεχνολογία. Όμως πιστεύω πως είναι βασικό να παραμείνουμε μπροστά. Στι ε, τεχνολογίες αυτές, ακριβώς για χάρη της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόληση Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε και με άλλους τομείς, με την πρωτοβουλία των Καθαρό Ουρανό ας πούμε, και με διάφορους ε, άλλους φορείς, με τους σιδηροδρόμους μεταξύ άλλων, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να, να συμπληρώσει ο ένας τις ανάγκες του άλλου και να μην πηγαίνει τίποτα, καμία προσπάθεια χαμένη. Το σημαντικό όμως ε, για τον τομέα αυτόν είναι ο συντονισμός. Ο συντονισμός γινόταν μέχρι τώρα μέσω των κοινών επιχειρήσεων. Είχαμε 11 συνολικά project, όμως ε, τώρα έχουν αυξηθεί ανάγκες ε, για το υδρογόνο ανεβαίνει σαν τεχνολογία και θα χρειαστεί καλό συντονισμός. Θεωρώ πως οι κοινέ επιχειρήσει θα πρέπει να είναι μια ενιαία ε, αφετηρία, μια ενιαία λύση. Επίσης, χρειάζεται να συνεισφέρουν όλοι μέσω ενός ε, κομβικού σημείου ε, μετάδοσης γνώσεων για το υδρογόνο. Τέλος, θεωρούμε πως θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε διαφορετικά ποσοστά χρηματοδότησης ανάλογα με τις ανάγκες μας. Και τέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα μέσα για τον επιτυχημένο συντονισμό. Και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και επιχορηγήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Εταιρικέ σχέσει και συμπράξεις δημοσίου-δημοσίου. Ε, Τώρα το λόγο έχει ο, ο κύριος ε, Νίντερλάντερ ε, σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση για την υποβοηθούμενη Ζωή, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε εδώ για τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από το πρόγραμμά μας και τη διαδικασία από εδώ και πέρα. Το πρόγραμμά μας λοιπόν πρόκειται για μια διεθνή εταιρική σχέση δημοσίου-δημοσίου. Έχουμε ε, ε, πάνω από 20 μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέχρι την Ταϊβάν. Ε, Έχουμε να κάνουμε με την τεχνολογία, και καινοτομία, υποδομές ε, και περιφερική φορείς. Πρόκειται για έναν διαθεματικό, διατομιακό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά και τη δημογραφική αλλαγή. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε πώς η Ευρώπη μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης ε, των ηλικιωμένων. κοιτάζοντας ε, τις ε, δημογραφικές τάσεις τα επόμενα 10-20 χρόνια. Είχαμε την έκθεση του ΩΣΑ, έκθεση ΣΑΠΗΡ για το μέλλον, που δείχνουν ότι πρέπει να λάβουμε δράση βεβαίως έτσι συμβάλλουμε και στην βιωσιμότητα του υγειονομικού συστήματος, συστήματος περίθαλψης, αφαιρώντας κάποια πίεση από τις υποδομές μας, καθώς θα ε, γυράσκει ο πληθυσμό, είναι και μια οικονομική δυνατότητα να έχουμε ένα νέο ευρωπαϊκό age H-Tech, που θα συνδέεται και με τον τομέα της πληροφορικής Έχουμε μια δεκαετή εμπειρία ε, με τη συνεργασία με δημόσιους χρηματοδότες και εμπλεκόμενα μέρη που είναι τελικοί χρήστες, σύλλογοι ηλικιωμένων ή και ευγυρίας και νοσοκομεία για να έχουμε μια καινοτομία φιλική προς ε, ε, τους ε, για να δούμε πώς μπορούν οι άνθρωποι να μένουν περισσότερο στο σπίτι τους, ασφαλείς, ε, κοινωνικά δικτυωμένοι και πώς θα διατηρήσουν και τις φυσικές τους ε, ικανότητες. Βέβαια όλα αυτά είναι, παίρνουν χρόνο για να φτάσουν στην αγορά. Από το 2008 μέχρι το 2013 εξετάσαμε ένα δείγμα 50 ε, έργων από τα 150 και τα 20 από αυτά έφεραν λύσεις στην αγορά. Πρόκειται για μια αναδυόμενη και αναπτυσσόμενη αγορά. Ταυτόχρονα, είπατε και εσείς πρέπει να, να είμαστε κοντά στους πολίτες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο οικοσύστημα. Δεν μιλούμε για το εθνικό επίπεδο. Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα εργαστούμε και μέσω προγραμμάτων ε, που ε, βρίσκονται σε έτσι, τοπικό επίπεδο και μεταξύ χωρών σε τομεί που έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Τρίτον, θέλουμε και θεσμικό κεφάλαιο πλέον. Δεν είναι απλή διαδικασία ε, αυτή της δημόσιας χρηματοδότησης όταν έχουμε διάφορους δημοσιονομικούς περιορισμούς και διαφορετικά μέτρα ε, σε κάθε χώρα και ταυτόχρονα έχουμε και αποκεντρωμένο σύστημα και παράλληλα δημοκρατική διακυβέρνηση, γιατί όλοι αυτοί οι δημόσιοι φορείς συνεργάζονται ε, σε έναν φορέα όπου υπάρχει και συνέλευση και ε, συμβούλιο ε, και οι δημόσιοι φορείς γενικά δεν έχουν συνηθίσει μια τέτοια προσέγγιση. Η δημογραφική αλλαγή είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ηλικιωμένους, έχει να κάνει με όλους τους πολίτες. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με μια σειρά άλλων εταιρικών σχέσεων ε, του ορίζοντα 2020, το 2REACH, το JPI MYBL, EIP στο AHA και του καθεξής. γιατί υπάρχουν και διαφορετικές αρμοδιότητες ε, σε κάθε τομέα. Υπάρχουν ήδη εμπειρίες και διαδικασίες και υποδομές. Δεν χρειάζεται να τα επανεφεύρουμε όλα αυτά. Θέλω μια εταιρική σχέση που πραγματικά αφορά το τομέα της υγείας. Αν δείτε την, ε, το θέμα της γύρανσης, έχουμε να κάνουμε με την πρόληψη, και με άλλους τομείς, έρευνα, καινοτομία, όλα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν για ένα καλύτερο ε, πλαίσιο πολιτικής ε, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, από κοινού και με την τεχνολογία και την οργανωτική καινοτομία. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία λοιπόν. Χρειαζόμαστε και άλλα επιχειρηματικά μοντέλα και άλλα μοντέλα οργάνωσης. Και βέβαια πάντα σε περιφερειακό επίπεδο να δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα για απορρόφηση των νέων προτάσεών μας. Πρόκειται για μια εταιρική σχέση χρηματοδότησης. Κλείνοντας, σαφώς και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και θέλουμε και τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη δημογραφική αλλαγή με την κλιματική αλλαγή. Μίλησε για την πράσινη συμφωνία. Καλό είναι να έχουμε και μια ε, συμφωνία μεταξύ γενεών. Γιατί και πάλι μιλούμε για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε την εκπαίδευση να αξιοποιήσουμε ε, στο έπακρον τις υποδομές μας, να βρούμε νέους τρόπους να ε, κάπως ε, να ελαφρύνουμε την πίεση στις υποδομές περίθαλψης και χρειαζόμαστε και νέες υποδομές. Πιο, πιο κοντά στον πολίτη, με βάση την κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας, για Νίντερλάντε. Μας εξήγησατε πώς, ε, τι δουλειά κάνετε και τελευταία, αλλά σημαντική, να μας εξηγήσει την ε, εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, την ε, κυρία Άντζελ Σορντούνια, εξελιχτική διευθύντρια του ΣΠΑΙΡ, εταιρική σχέση Το Spire είναι μια εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα που έχει μια συστημική προσέγγιση που βοηθάει την κοινωνία, δεν μπορεί να το κάνει κανένας πολίτης μόνος του. Εκπροσωπούμε 8 τομείς, 900 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ. Ε, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τζίρος. Έχουν μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, συγγνώμη, ε, και έχουμε μια μοναδική συνεργασία που δεν έχει ξανακινήσει στην Ευρώπη. Έχει δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνη σε διάφορου τομεί μεταξύ διάφορων, διάφορων τομέων που συνετέχουν στο ΣΠΑΙΡ. Έχουμε 150 μέλη αυτή τη στιγμή που ε, είναι από περιφέρειες, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, ε, διάφορα είδη μελών έχουμε εταιρείε βέβαια. Είμαστε σε 20 χώρες αυτή τη στιγμή παρόντες και το 95% των επενδύσεών μας ε, γίνονται ε, σε προϊόντα στην Ευρώπη. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα προγράμματα του ορίζοντα. Είμαστε τμήμα το, της αλυσίδας αξιών των εταιρικών σχέσεων στην αρχή έχουμε εταιρικέ σχέσεις πάνω-πάνω ε, EIT για, τα, για τις πρώτες ύλες. Ε, εμείς είμαστε στο μέσο της αλυσίδας και στο τελικό κομμάτι της αλυσίδας. Έχουμε μοναδική θέση σε αυτή την εταιρική σχέση, γιατί η μείωση των εκπομπών διοξείδου του άνθρακα στη μεταποιητική βιομηχανία θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα. Ε, οτιδήποτε συμβεί στα προϊόντα, οποιαδήποτε εξοικονόμηση διοξείδου του άνθρακα θα φτάσει ως τις πόλεις και θα πάμε πίσω, θα κλείσουμε το βρόχο, θα χρησιμοποιήσουμε όλους αυτούς τους πόρους, ε, θα τους ξαναβάλουμε στο βιομηχανικό process, στη βιομηχανική διαδικασία ε, και θα υλοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο το όραμα ή θα συνεισφέρουμε στην υλοποίηση του όραματος της Προέδρου Φόντερ Λάιεν. Είμαστε μια νέα εταιρική σχέση. Ξεκινήσαμε το 2014, ε, αλλά δείχνουμε ήδη ότι έχουμε σημαντική επίπτωση για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Μέχρι το τέλος του 2018 είχαμε 89 έργα. Ε, παράγοντας μόχλευση 8,5%, 4,5% δισεκατομμύρια επενδύσεις έχει πολλά ε, νέα συστήματα και τεχνολογίες, πολλές είναι καινοτόμε. Αυτά τα έργα θέτουν τη βάση για να καθορίσουμε μια νέα στρατηγική για το Spire. Ε, στους περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους πάμε πολύ καλά. Μείωση των, συμπεριλαμβάνουμε εδώ την ε, μείωση, την μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, αύξηση των ε, ανέωσιμων πηγών ενέργεια, ε, μείωση των αποβλήτων. Ε, μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα του στόχου μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Το δουλεύουμε αυτό, αλλά χρειάζεται πραγματική στήριξη για να, πραγματικά, να, για να ειδοποιήσουν πραγματικά του στόχου του Green Deal. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που συμμετέχουν στο Spire ε, τα πάνε καλύτερα από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 28. Έχουν περισσότερε θέσει απασχόληση ή περισσότερου νέου εργαζόμενου από τι ε, υπόλοιπε εταιρείε έχουν υπερδιπλάσιο τζίρο από τις υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στο τα λοιπά. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα δικό χάρτη με βάση την, το όραμά μας και κάνουμε μια πρόταση. Ξέρουμε ότι για την κλιματική ουδετερότητα και την ε, κυκλική οικονομία ε, πρέπει να τροποποιήσουμε την ε, μεταποιητική βιομηχανία, να μειώσουμε τις ε, προβληματικές ε, τεχνολογίες. Η πρότασή μας για την αξία είναι να δημιουργήσουμε μια διαδικασία, μια βιομηχανία μεταποίησης άμεση, ψηφιοποιημένη, που θα υλοποιεί τους στόχους του Green Deal. Έχουμε τις εξής φιλοδοξίες. Να κλείσουμε καταρχάς το τεχνολογικό χάσμα, ε, του 2050 είναι να χρησιμοποιήσουμε τους κυκλικούς πόρους για σχεδόν μηδενικά απόβλητα στις χωματερές και μηδενικά λίματα σχεδόν. Επίσης πρέπει να έχουμε ε, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Αν δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει αυτή, ε, ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο θα εξαφανιστούμε. Και έχουμε μοχλούς μετασχηματισμού. Έχουμε τέσσερι τέτοιου μοχλού, 16 τομεί ε, καινοτομία, 36 προγράμματα καινοτομία. Δεν θα επεκταθώ, δεν έχω χρόνο. Θα μιλήσω για τα κέντρα κυκλικότητας, Hubs for Circularity. Όταν ε, ετοιμάσαμε το όραμά μα ήρθαν σε επαφή μαζί μας οι περιφέρειες και εδώ συνδεδόμαστε πολύ καλά με την ιδέα για τις κλιματικά ουδέτερε πόλεις και τις, ε, τη μείωση των εκπομπών. Με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε λοιπόν με τις περιφέρειες και αυτό που θέλουμε από τις περιφέρειες είναι να συνέλθουν όλοι οι φορεί των περιφερειών και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο με δεσμεύσει με ένα πρόγραμμα επενδύσεων να δούμε τις ανάγκες και τη ζήτηση αυτής της περιφέρειας και της κοινωνίας της περιφέρειας αυτής και βρίσκει λύσεις μέσω έρευνας και κοινοτομία ή μέσω άλλων μέσων για να το πετύχουμε αυτό. Και να υπάρξει συνεργασία με άλλους εταίρους από τις άλλες αποστολές. Επίσης, δημιουργούμε και αυτά τα λεγόμενα marbles. Δεν υπάρχει επίπτωση εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη προϊόντων. Ε, πρέπει να ξεπεράσουμε τον ορίζοντα Ευρώπη, να έχουμε αυτά τα μεγάλα προγράμματα επίδειξης, ε, μεγάλης κλίμακας, ούτως ώστε να φανεί ότι υπάρχει επίπτωση. Στο οδικό μας χάρτη έχουμε προβλέψει τις ανάγκες, ε, τις επενδυτικές ανάγκες ε, ύψους 70 δις για να δούμε ε, τι προγράμματα επίδειξης έχουμε ανάγκη για να τα αναπτύξουμε. Το Spire συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά αντιμετωπίζει κινδύνους σε ό,τι αφορά τι μακροπρόθεσμε επενδύσεις. Ε, συμμετέχουμε σε κάποια από τα κλάστερ του ορίζοντα Ευρώπη και κατά την άποψή μα αυτό είναι σημαντικό. Το προπολογισμό του ορίζοντα Ευρώπη να είναι πάνω από τα 100 δις. Και πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει στήριξη για την καινοτομία, η οποία να μην έχει άνωτατο όριο. Τέλος. Είμαστε έτοιμοι ως νέος ε, εταίρος να έχουμε μια υψηλότερη φιλοδοξία. Έχουμε νέους ε, φορείς στην εταιρική μας σχέση πρόσφατα. Έχουν έρθει εταιρείε πληροφορική, ε, ΜΚΟ, σε επαφή μαζί μας. Είμαστε σε συζήτηση για να δούμε ποιοι νέοι ας πούμε, τομείς και φορείς θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Spire. Και έχουμε βάλει στις συζητήσεις πάνω από 100 εκπροσώπους από ΜΚΟ, τη βιομηχανία, τα μέλη και μη μέλη του Spire, κράτη-μέλη, ε, περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών. Δύο λεπτά για τον εισηγητή, ενάμιση λεπτό για τους σκιώδεις και ένα για τους υπόλοιπους. Και θα δούμε μετά πώς θα χωρίσουμε το χρόνο για τις απαντήσεις. Ξεκινάμε από τον κύριο Νίκα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να χαιρετήσω ε, τις εισηγήσει ε, των ομιλητών μας. Ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Το πρώτο ερώτημα Εφόσον δεν έχουμε ακόμα τελικό προπολογισμό για την επόμενη πραγματική περίοδο, πώς εσείς προγραμματίζετε τις ε, δραστηριότητές σας ε, για τους στόχους ε, των εταιρικών σχέσεων που έχετε παρουσιάσει σήμερα. Για το Clear Sky. Στη σχέση με την αρχική εταιρική σχέση της πραγματικής περίοδου 7, έχετε καινούργια στοιχεία. Θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Μπεϊβούκ. Ε, για τις ε, κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο. Είπατε ότι η παραγωγή γιγαβάτ ε, θα πρέπει να προχωρήσει. Πότε θα γίνει αυτό. Μετά σήμερα μιλήσαμε πολύ για υδρογόνο. Κάποιοι είπαν ότι η παραγωγή υδρογόνου είναι πολύ ακριβή, άλλοι λένε ότι η παραγωγή αυτή δεν είναι εφικτή, γιατί καταναλώνουν πολλή ενέργεια και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Πότε όμως θα υπάρχει μια τέτοια τεχνολογία με βάση γιγαβάτ που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλη κλίμακα και πότε θα είναι έτοιμη μια τέτοια τεχνολογία δεν έχουμε επαρκείς ε, δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Χρειαζόμαστε λοιπόν να, και πρέπει να ε, διερευνήσουμε όλες τις εφιστάμενες τεχνολογίες. Το υδρογόνο είναι μια σημαντική τεχνολογία και θα ήθελα συνάδελφοι να ακούσουν ε, τι απαντήσεις σας. Για το Spire. Μόνο τρία μέλη είναι από την Ανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβενία. Στο πλαίσιο του Spire, οι περισσότερε επιχειρήσει έχουν ε, έρθει μέσα στις χώρες Ανατολική Ευρώπης, αλλά δεν ε, υφίστανται εκεί. Η Ανατολική Ευρώπη λέμε ότι θα ε, παράγει βιομάζα και ενέργεια από βιομάζα και τα εργαστήρια θα πρέπει, όμως βλέπουμε ότι θα είναι στη Δυτική Ευρώπη. Ε, τώρα μιλάμε για προγράμματα που είναι από το 1964. Η Σοβιετική Ένωση ε, μας παρουσίαζε τα έργα και εμείς δίναμε τις πρώτες ύλε στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτή η πρόταση δεν ε, θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορούν αυτοί να είναι οι στόχοι μας για το 2050. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλλερ. Κάτι πιο γενικό θα πω. Βλέπουμε ότι έχουμε την Πράσινη Συμφωνία και απέναντί τη μια πληθώρα μέσων και προγραμμάτων. Οπότε νομίζω πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θεωρώ λοιπόν ότι Πρέπει να καταβάλουμε μια συλλογική προσπάθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Αν δείτε τις συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου φορέα, θα παρατηρήσετε ότι ποτέ δεν συμπεριλήφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. στο... Υπάρχει συμμετοχή των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 185, όμως ε, η πολιτική δεν χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία και δεν τα εντάσσει στο πολιτικό εξάμεινο. Ούτε μία αναφορά δεν υπάρχει στα αποτελέσματα του άρθρου 185. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να σπαταλάμε χρήματα και να υπάρχει κατακαιρματισμός. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω ποιε είναι και οι προσδοκίες σας από το Συμβούλιο το οποίο χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τώρα για τη συμπράξη του άρθρου 87. Τι περιμένετε να γίνει μετά το Brexit. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, αγοράς ε, η, αεροπορική βιομηχανία. Το Ενωμένο Βασίλειο συμμετέχει στην κοινοπραξία της Airbus, οπότε τι θα γίνει μετά την αποχώρησή του. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές ε, αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ οι οποίες θα γίνουν πελάτες αυτής της νέας τεχνολογίας. Ποιο θα είναι λοιπόν, λοιπόν ο αντίκτυπος του Brexit στο καθαρό ουρανό. Και τελευταία ερώτηση πιο πρακτική. Σε σχέση με το υδρογόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς το υδρογόνο συμμετέχει σε αυτήν την αλυσίδα αξία. Τώρα βρίσκεται εκτός προγράμματο κινητικότητας, παρά το γεγονό ότι στην, ε, στον τομέα αυτό μπορείς ε, να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα χρησιμοποιώντα υδρογόνο. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικό και οι τιμές του υδρογόνου επηρεάζονται εύκολα. Ποιο είναι λοιπόν το σκεπτικό για το υδρογόνο πέρα από αυτό, πέρα από την προσέγγιση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έλερ, κυρία Τζαμπάλεβα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες για αυτό το θέμα. Αλλά θα περιοριστώ λοιπόν. Και εγώ την ίδια ερώτηση με τον κύριο Έλερ έχω. Τι θα γίνει δηλαδή μετά τον Brexit. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι δικέ σας προσδοκίε και τι μπορεί να αλλάξει. Βέβαια ξέρω ότι και εσείς από εμά περιμένετε, οπότε ο καθένας κάποιον περιμένει. Αλλά τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Ήμουν ε, η συγγήτρια για τις ε, σχετικές απαλλαγές στο Κοινοβούλιο και έχω μια εικόνα του πώς έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια. Γι' αυτό μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του Καθαρού Ουρανού. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η επιτυχία της ε, εταιρική σας σχέσης και το φιλόδοξο σχέδιο που έχετε. <clears throat> Η αεροπορία πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό κομμάτι της μελλοντική βιομηχανικής μας πολιτικής. Νομίζω ότι ο καθαρό νόσο είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Στην Τσεχία το είδα με τα μάτια μου πόσο επιτυχημένο ήταν. Χρειαζόμαστε όμως μια ξεκάθαρη στρατηγική. Και στην Επιτροπή μας πρέπει να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε αυτή την πρόσθετη χρηματοδότηση, διότι αν δεν φτάνει η χρηματοδότηση υπό τον πυλώνα 2, υπό την ε, δέσμη δηλαδή της κινητικότητας θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο χρηματοδότησης ή ίσως υπό τον πυλώνα της ε, βιομηχανίας ή να βρούμε συνέργειες για να το επιτύχουμε. Νομίζω πως οι συνέργειες είναι η λέξη κλειδί εδώ. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να δούμε τις συνέργειες μεταξύ όλων των ε, μόρφων εταιρικών σχέσεων, όλων των συνεργασιών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρατρύνω να ενισχύσετε τις συνέργειες ε, μεταξύ των, του προγράμματος Καθαρός Ουρανός, Καθαρός Ουρανός 2, μια που υπάρχει και πρώτερη εμπειρία. Τι γνώμη έχετε λοιπόν για τις συνέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίτση. Μας καθησυχάσατε με τα λόγια σας κύριε Διευθυντά, κύριε Κλάιν αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το clean sky, για τους καθαρούς ε, ουρανούς. Γιατί δεν είναι ανοιχτό σε όλους αυτό, αυτή η εταιρική σχέση. Δηλαδή χρηματοδοτούνται μόνο λίγες και τεράστιες επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες αποκλείονται. Λίγες, ε, λίγες, ε, λίγα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα συμμετείχαν και μόνο 420 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλα τα 28 κράτη-μέλη. Ε, η συνεργασία ε, μεγάλων επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί αντιπεραιτέρω για να είναι βιώσιμος ο κλάδος. Δεν πιστεύετε ότι η καθαρή ουρανή θα μπορούσε να είναι πραγματικό εργαστήρι για να δημιουργήσει και να ενισχύσει αριστεία διασυνοριακού χαρακτήρα. Αυτή είναι η ερώτηση για τον κύριο Νίντερλάντερ και Ορντούνια είπατε ότι είσαστε παρόντες σε 19 και 20 ε, χώρες ο ένας και ο άλλος. Ε, πώς, θα, πώς θα προσπαθήσετε για να μην αφήσετε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός, να τις, μετά, να τις συμπεριλάβατε όλες. Επίσης, αν δεν ξεκινήσουν μαζί όλες οι αποστολές, όπως εμείς θεωρούμε, δεν θα γίνει. Πώς θα υπάρχει ευθυγράμμιση με τους στόχους των εκπομπών ε, σε όλα τα επίπεδα γιατί ε, παίρνουν αυτές οι αποστολές σχεδόν το μισό του προπολογισμού του δεύτερου πυλώνα. Ε, πώς θα συνεργαστείτε διάφορες επιλογές, θα κάνετε συνεδριάσεις, πώς θα επικοινωνείτε για να μην έχετε επικαλύψεις. Ευχαριστώ. Είστε το Το Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα μόνο για τους ε, καθαρούς εθέρες. Βλέπουμε ότι παγκόσμια αυξάνονται οι αεροπορικές μεταφορές και στην Ευρώπη και αν ε, σε βάθος χρόνου μιλούμε για διπλασιασμό των αερομεταφορών... μεταφορών και από την άλλη έχουμε και δέσμευση μείωση των εκπομπών ε, για να παραμείνουμε μάλλον στα σημερινά επίπεδα εκπομπών θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες, υφιστάμενες τεχνολογίες για να περικόψουμε τις εκπομπές κατά 50%. Είναι εφικτό αυτό. Μπορούμε όντως να περιορίσουμε τόσο δραστικά τις εκπομπές χωρίς ε, να υπάρξει κάποια τρομερή νέα ε, τεχνολογία όσης. Δεν ξέρω αν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων τεχνολογιών μας επιτρέπουν ε, κάτι τέτοιο ή αυτό θα έχει αντίκτυπο στις ε, τιμές των καυσίμων. Εάν δεν ε, μπορούμε να βασιστούμε σε κάποια νέα καταπληκτική τεχνολογία την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε. Τρεις παρεμβάσεις. Η κυρία Καρβάλιο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Για τις κοινέ επιχειρήσεις, ε, ένα στο ερώτημα. Αερονεφυγική και υδρογόνο. Μαζί και με την παρουσίαση των έργων. Νομίζω ότι έτσι με αυτό το νέο κύκλο συνεργασιών θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Και χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια. Και αυτό θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη προβολή των έργων. Είπατε ότι υπάρχουν πολλοί εταίροι, αλλά σε κάποια κρατημέλη τα, τα προγράμματα ακόμα δεν είναι γνωστά πρέπει να υπάρχει και καλύτερη κατανομή, γιατί έχουμε πολύ καλούς εταίρους σε όλη την Ευρώπη που δεν γνωρίζουν αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Thank you, thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε, κύριο Ιζάμπς. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείται. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την ε, αναδιοργάνωση του πλαισίου εταιρική σχέσης που θα ξεκινήσει με το επόμενο πι. Το 2017 η Εστονική Προεδρία ε, δημοσίευσε μια έκθεση για τις ευρωπαϊκές εταιρικέ σχέσεις ε, όπου εντόπιζε ορισμένες αδυναμίες της υφιστάμενης δομής. Κατακαιρματισμός, έλλειψη εμπλοκής των κρατών μελών στην ε, θέσπιση ορισμένων KPIs. σε φορά την ε, συλλογή και παρακολούθηση των ε, δεδομένων. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα από την ε, πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει κάποια δυνατότητα περαιτέρω βελτίωση. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπλός από τους πλασίνους. Ευχαριστούμε πολύ. Υπήρξε μια αναθεώρηση προγράμματος ε, το 2017. Ποιες ε, ήταν ε, οι βασικές παρατηρήσεις σας με βάση αυτή την αναθεώρηση. Προτείνετε κάποιες προσαρμογές εν ώψη και της Πράσινης Συμφωνίας και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας εν ώψη του 2050. Ποιο συγκεκριμένα για, το υδρο... την εταιρική σχέση για το υδρογόνο. το πλήρες ανανεώσιμο υδρογόνο το λαμβάνετε υπόψη σας στο, πρόγραμμά σας. Μιλήστε για το 24% των συνολικών ε, της συνολικής ζήτησης ε, ε, ενέργειας από το υδρογόνο. Αυτό πάλι πρόκειται για πλήρως ανανεώσιμο. Και θα ήθελα να συζητήσουμε με τον κύριο Έλλας πόσο υδρογόνο χρειάζεται η βιομηχανία. Γνωρίζουμε ότι για να αντικαταστήσουμε το υδρογόνο στην χημική βιομηχανία <coughs> Ε, θα, πάρει καιρό. Κάτι τελευταίο, διαφάνεια λέγατε. Κάποιοι θέλουν να δουν ποιοι είναι οι εταίροι, ποιες είναι οι ΜΚΟ και στο, στους αυτό δεν είναι σαφές. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη να υπάρχει διαφάνεια για τους πολίτες. Και κάτι τελευταίο, διακόπτε Πρόεδρος, για τη γραμματεία. δεν ε, φαίνονται οι διαφάνειες από τις οθόνες. Ειδικά αν κάθεται κάποιος πίσω-πίσω ε, στην αίθουσα. Ευχαριστούμε κύριε Μπλουμ. Ναι, θα δούμε πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τις τεχνικές εγκαταστάσεις και στους ιστοτόπους βεβαίως θα βρείτε τις παρουσιάσεις αυτές. Παρακαλούμε να μας τις στείλετε. Δυόμιση λεπτά έκαστος. Να αναφέρω ότι στις 12.30 θα σταματήσει η διερμηνία, γιατί ξεκινήσαμε πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς και θα συνεχίσουμε στα αγγλικά μετά από τις 12.30. Δυόμιση λεπτά ο καθομιλητής λοιπόν. Ας ε, ξεκινήσουμε αντιστρόφως ξεκινώντας από την κυρία Ορντούνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Πρώτον, παρουσία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το Spire σαφώς και έχει μεγαλύτερη παρουσία σε χώρες όπου ο κλάδος της μεταποίησης είναι πιο ε, διαδεδομένος, ειδικά εκεί που εδρεύουν αυτές οι επιχειρήσεις. Σίγουρα υπάρχουν και τις επιχειρήσεις σε άλλες χώρες που δεν, και δεν υπάρχουν στο Μητρό μας. Συνεργαζόμαστε ιδιαίτερως με τις χώρες ε, τις ανατολικές. Με την Πολωνία συναντιόμαστε συνήθως μία φορά το χρόνο. Ε, Λιθουανία τώρα. Ε, ε, ε, είμαστε σε συζητήσεις και με τη Λιθουανία και με άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για να βρούμε περισσότερα ενδιαφέρμενα μέρη από εκεί. Οργανώνουμε στοχευμένες εκδηλώσεις, συναντήσεις. Πάντα έχουμε και άλλες συναντήσεις στο περιθώριο δηλαδή. Και με τους κόμβους κυκλικότητας ε, αναμένουμε αυτό να ενισχυθεί. Ο κατάλογος των μελών μας ε, είναι δημοσιευμένος στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να τον δείτε εκεί. Να, εκεί θα δείτε και τη ΜΚΟ και όλα μας τα μέλη. Μετά, ε, εμείς εργαζόμαστε μέσω ομάδων εργασίας που είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για την ε, συλλογή πληροφοριών και απόψεων ε, και με ευρωβουλευτές, συζητήσεις με ευρωβουλευτές για να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις και εδώ με τις κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο, τα συζητήσαμε όλα και με το BBI από πλευράς αξίας περισσότερο, αλλά είναι σαφές ότι και η βιομάζα ε, αποτελεί τμήμα του Spire. Η βιομάζα είναι μια τέτοια πηγή, ενώ και το PPI οτιδήποτε δεν είναι αξία δεν εμπίπτει στα πεδία εφαρμογή. Σημαντικό είναι να υπάρχουν δημόσιες διαβουλεύσεις με διάφορες μορφές εμπλεκομένων ε, μερών, διάφοροι κλάδοι, ε, κοινότητα των πολιτών και το καθεξής. Για το Brexit, κλείνοντας, σίγουρα θα μας επηρεάσει όλους. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα εξαρτηθεί από την ε, τελική συμφωνία, αν γίνουν ε, συνδεδεμένη χώρα για τον ορίζοντα, για εμάς τα πράγματα θα συνεχίσουν όσο έχουν. Όπω και με όλε τι υπόλοιπε συνδεδεμένε χώρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σίντριλάντερ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα πω ε, την άποψή μου για τον Brexit. Χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστέ, λοιπόν. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του Μόνο Βασιλείου δεν συγχρηματοδοτεί προγράμματα, θέλει όμω να παραμείνει συνδεδεμένη μαζί μα. γι' αυτό λοιπόν θα διατηρήσουμε αυτή τη σύνδεση. Το, η επιχειρήση του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμα συνδέονται με τις δραστηριότητές μας, οπότε περιμένουμε μέχρι να καταλαγιάσει λίγο ο πολιτικός αυτός θόρυβος και να δούμε πώς μπορούμε να τις εντάξουμε, ίσως όπως ε, γίνεται και με την ε, Νορβηγία ή την Ελβετία, τον Καναδά. Τώρα, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία Βορρά Νότου Ανατολής Δύσης και συνεργαζόμαστε και με άλλες μορφές εταιρικών σχέσεων έτσι ώστε να ε, συγχωνευτούν και να δημιουργηθεί μια νέα μορφή εταιρική σχέση η οποία θα αυξήσει το πεδίο δράσης μας. Υπάρχει και η ομάδα εργασίας των κρατών μελών με πάνω από 50 μέλη. Υπάρχουν και άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτές ε, τις ε, ομάδες, οπότε νομίζω πως η κάλυψη είναι αρκετά καλή και θα βελτιωθεί στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση ναι, είναι όντω πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά δίνεται έμφαση στην πράσινη συμφωνία, αλλά σίγουρα είναι εθνική αρμοδιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, διότι η δημοκρατική αλλαγή μας αφορά όλους στην Ευρώπη. Και πρέπει να συνδεθεί με την έρευνα και την καινοτομία με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να συνεργαστούμε με άλλες μορφές εταιρικέ σχέσεις ή με τους μεγάλους εταίρους μας από τον κλάδο της βιομηχανίας. Φυσικά αυτό γίνεται καλή πίστη, αλλά αν δεν δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δεν θα αποφύγουμε αυτές τις επικαλύψεις. Ε,